Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να αρχίσουμε. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα το απόγευμα είναι η έκθεση Τάραντ για το ρόλο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας σε περισσότερες περιπτώσεις κρίσεων που φύλλονται στο κλίμα και στις φυσικές καταστροφές. Πρόκειται για γνωμοδότηση πρωτοβουλία της Επιτροπής μας. Στην πρώτη συζήτηση που έγινε στην 21η Ιουνίου, φάνηκε ότι οι περισσότερες πολιτικές ομάδες αναγνώρισαν πόσο σημαντικές ε, απειλές, πόσο σημαντική είναι η απειλή για την ασφάλεια εξαιτία των κλιματικών αλλαγών και των φυσικών καταστροφών και είπαν ότι θα πρέπει οι δυνατότητες και οι προσαρμογές της ΚΕΠΑ να γίνουν για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε αποδοτικά. Δεν υπήρχε όμως συμφωνία, υπήρχε κάποιο σκεπτικισμό όσον αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα που προτάθηκαν. Γι' αυτό αποφασίσαμε να οργανώσουμε σήμερα μία ε, ακρόαση με τους εμπειρογνώμενες για να βοηθηθούμε. Έχει παρατεθεί προς μια κατάθεση τροπολογιών μέχρι την Παρασκευή 13 για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να λάβουν υπόψη τις συζητήσεις που θα γίνουν. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τώρα τους εμπειρογνώμενους και να τους ευχαριστήσω το ενδιαφέρον και τον χρόνο που μας αφιερώνουν. Πρώτα απ' όλα έχουμε μαζί μας τον υπονάβαρχο Νέιλ Μωρισέτη, εντεταλμένο για θέματα κλίματος και ενεργειακής ασφάλειας του Υπουργείου Άμυνας και Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου έχουμε τον υπονόμορφο Bruce Williams, πληρωτή Γενικό Διευθυντή του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον, Graham, τον Christian ο Διευθυντή της ε, Ευρωπαϊκού Υπηρεσίας Άμυνας και τον Τόμ Σπένσερ, Αντιπρόεδρο, Γενικό Συμβουλευτικό Στρατιωτικό σύμβουλο και πρώην Ευρωβουλευτή. Πριν να δώσω το λόγο στους συναδέλφους της ε, εμπειρογνώμονες θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Τάρατ να μας κάνει μία μικρή εισαγωγή στο θέμα. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που μπορεί να λάβει σήμερα χώρα αυτή η συνάντηση με τους εμπειρογνώμενους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ντονζόν και τον κύριο Παλέτσκι που έκαναν, ε, οργάνωσαν αυτή την ε, συνάντηση. Είχαμε πολλές συναντήσεις ήδη με τους κοιόδης ηγητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων καθώς και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εξωτερικής Υπηρεσίας, της, Γενική της Γενικής Διεύθυνσης Πόσο τα Κλιματολογικά και με εκπροσώπους ε, εξωτερικούς και μπόρεσα έτσι να φτιάξω την εκθεσή μου προσπαθώντας τα σχόλιά μου να πηχούν τι απόψει των διαφόρων που συμμετείχουν σε αυτέ τι συντηρήσει, θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να σα πω ότι το σημείο κίνηση αυτή τη έκθεση είναι το άρθρο 41.3 έως 5 της Συνθήκης Λισαβόνας που αναφέρει πολλά χρήσιμα σημεία τα οποία δεν έχουμε αναπτύξει όπως θα έπρεπε και πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να επωφεληθούμε από όλες ευκαιρίες που μας προσφέρει η συνθήκη. Σήμερα θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το πράγμα, αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας που αφορά την ε, κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σφαιρικά στην ε, ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και πώς στα πλαίσια της ΚΕΠΑ θα κάνουμε κάτι. Προσπάθησα προσεκτικά στην έκθεση αυτή να μην κάνω επικαλύψεις, όπως ανέφερα οποιαδήποτε δράση είναι επικάλυψη δεν θα πρέπει να είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε. Δεν θα πρέπει να κατασπαταλώνονται οι πόροι. Αναγνωρίζουμε τι έχει κάνει η Επιτροπή και επίσης η εξωτερική υπηρεσία. Αλλά προσπαθούμε παρόλα αυτά να τους δώσουμε ένα νέο λόγο ύπαρξης. Βεβαίως, οι μηχανισμοί προστασίας των ε, πολιτικής προστασίας δεν μπορώ να πω ότι είναι εκτός όλων αυτών των μηχανισμών. Παρά το γεγονός ότι ασχολούμεθα μόνο με την ΚΕΠΑ, πρέπει να πω ότι αναγνωρίζουμε την εργασία που έκανε η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και άλλοι που ε, συμμετέχουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε με την έκθεση αυτή είναι κυρίως τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα, ποια πολιτική θα ακολουθεί από την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων και ποιες προτάσεις θα γίνουν ώστε να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από τα κονδύλια που έχουμε. Το pull and share είναι κάτι το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και μας, προστατεύει μας την να από κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές, όπως και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι θα πρέπει και εδώ να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Η κλιματική ασφάλεια, αν θέλετε, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δομές που υπάρχουν και πώς θα μπορέσουμε όλοι μεταξύ μας να δημιουργήσουμε μία task force της οποίας θα ηγηθεί κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να εφαρμόσει όλες τις αρχές τις οποίες θέλουμε ώστε να έχουμε την κατάλληλη πολιτική στον τομέα αυτό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Όσοι με βοήθησαν και συνεισέφεραν ε, για τη σύνταξη του κειμένου τους ευχαριστώ και όσοι μας επέκριναν ας ακούσουν τι έχουμε να πούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους του πάνελ. Για να μας πείτε τις απόψεις σας. Έχετε περίπου 10 λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τη δική μας απόψη, η προοπτική αυτών των ζητημάτων βάσει τριών ετών ω εντεταλμένο του Ηνωμένου Βασιλείου για την ενέργεια και την ασφάλεια. Πιστεύω ότι αναγνωρίζετε όλο και περισσότερο τα τελευταία 5 και 10 χρόνια στον κόσμο ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, κοινωνικό ή οικονομικό ζήτημα, είναι όλα μαζί. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο έργο των Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στι πρωτεύουσε, Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένε Πολιτείε, ότι υπάρχουν ίσω συνέπειε. Ε, στην ασφάλεια και ειδικότερα στον τρίτο κόσμο. Θα επιστήσω την προσοχή σας, θα δώσω σε έναν χάρτη ώστε να σας ε, δείξω τι εννοώ. Οι επιπτώσεις ε, ανώδων των, ε, θερμοκρασιών του επίπεδου της θάλασσας αυτά μπορεί να επηρεάσουν τον κόσμο. Μπορεί να απολεστούν γιές, μέσα διαβίωσης, ε, μπορεί να επηρεάσει την ή και η άνοδος του επίπεδου των θαλασσών μπορεί να εξαφανίσει τα δέλτα ποταμών ε, στον Μπαγκλαντές ή σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτό μπορεί να υπάρξει σε περιοχές που ήδη υποφέρουν από πιέσεις, ελλείψεις ε, νερού, υπερπληθισμό, προβλήματα σύντησης, αυτό το επισημαίνεται στο χάρτη με τις σκιασμένες περιοχές ε, σε περιοχές της Κεντρικής Νότιας Αμερικής, Αφρικής, Ασίας, κοντά στο νησιμερινό, μια ε, ζώνη από την οποία διέρχονται και οι εμπορικέ οδοί. Η κλιματική αναλλαγή θεωρείται καταλήτης των απειλών, ε, ότι πολλαπλασιάζει τι απειλέ σε αυτές τι περιοχές. Αυτό που μας ανησυχεί εδώ στην Ευρώπη, που παρότι είμαστε ένα λευκό κομμάτι του χάρτη, δεν επηρεαζόμαστε άμεσα βραχυπρόθεσμα, αλλά το γεγονό ότι ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και εξαρτόμαστε από δραστηριότητες χιλιάδε μίλια μακριά μας, αυτή είναι η αιτία. Για παράδειγμα, ε, οι ακραίε καιρικέ συνθήκε στην Ταϊλάνδη πέρυσι επηρέασαν όχι μόνο την οικονομία της Ταϊλάνδης αλλά το γεγονός ότι κατασκευάζονται εξαρτήματα για αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν να ομολογηθούν σε άλλες χώρες και έτσι επηρεάζεται η γραμμή παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα. Επίσης ε, είδαμε ότι είχαμε έλλειψη σκληρών δίσκων για υπολογιστές επειδή εκεί κατασκευάζονται μικροτσίπ. Είμαστε σε έναν υψηλά παγκοσμιωμένο κόσμο και το ίδιο συμβαίνει και για την ενέργεια, η οποία διέρχεται από διάφορα κομμάτια, από διάφορα μέρη του κόσμου και έτσι η κίνδυνη είναι αυξημένη. Επίσης υπάρχει σχέση μεταξύ της έλλειψης τροφής, νερού και της κλιματικής αλλαγή. Εμείς χρειαζόμαστε βιώσιμες ε, συνεχείς ε, παροχές ώστε να εξασφαλίζεται η ευημερία και η ανάπτυξη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν γι' αυτό. Προτείνω να αναγνωρίσουμε τις επιπλέον επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να κατανοήσουμε τους κινδύνους. Και να το συγκρίνουμε με άλλες απειλές στην παγκόσμια σταθερότητα που ζήσαμε τον 20ο αιώνα. Μπορούμε να κατανοήσουμε πώς μπορεί να εκδηλωθούν και τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε αυτούς τους κινδύνους. Ε, προτεραιότητα δική μας πρέπει να είναι η μείωση αυτών των κινδύνων, σε ποια μέρη του κόσμου χρειάζεται δράση και με τη χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα απαιτήσει μια εξέλιξη των θεσμών από του εθνικού θεσμούς μέχρι τους διεθνείς, ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Για παράδειγμα, σε εθνικό επίπεδο ε, απαιτεί εθνική αντιμετώπιση και όχι τμηματική. Και σε διεθνές επίπεδο χρειάζεται τη συνεργασία πολλών οργανισμών για να επιτευχθεί αυτό. Ε, σε μια σύνοδο πέρυσι τον Ιούνιο στο Λονδίνο επισημάθηκαν διάφορα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη για δράση, χρειάζεται ανάγκη ηγεσία σε όλα τα επίπεδα. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική και τα στοιχεία κλιματική ασφάλεια πρέπει να έχουν συνοχή με την ευρύτερη κλιματική παγκόσμια στρατηγική. Πρέπει να ενισχύσουμε τι περιφερειακέ δραστηριότητε, αλλά να αποφύγουμε τι επικαλύψει μεταξύ θεσμών και δράσεων. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε νέου θεσμού, νέε επιτροπέ. Όχι. Χρειάζεται να διαβεβαιώσουμε ότι οι υπάρχουσε μπορούν να εξελιχθούν ώστε να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει. Και χρειαζόμαστε και ένα συγκεκριμένο σκεπτικό και διάλογο για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο τρόπο που αντιμετωπίσαμε αυτά τα ζητήματα, όπω είδα εγώ από τη δική μου θέση, ω εντεταλμένο για την ε, ασφάλεια τη ενέργεια, ε, εργάστηκα σε θέματα άμυνα, ε, στην υπηρεσία της κοινοπολιτείας είχα τρεις ρόλους χρειάζεται να κατανοήσουμε αυτά τα ζητήματα και να βεβαιώσουμε ότι υπάρχουν εθνικές στρατηγικές για αναγνώριση αυτών των προκλήσεων και ένταξή τους στο σκεπτικό των εθνικών στρατηγικών. Το είδαμε αυτό σε ορισμένες χώρες όπως το ΕΒ, Βασίλειο, στην Εθνική Στρατηγική για την Άμυνα για το 2010, αλλά και στην Αμερική σε παρόμοια στρατηγική το ίδιο έτος. Στη συνέχεια πρέπει να συνεργαστούμε με το, στρα... το στρατό ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να αποκτήσουμε τις ικανότητες και το τρίτο επίπεδο αποτελεί συνιστά την όλη κυβερνητική προσέγγιση ώστε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς. Δεν μιλάμε για μια συζήτηση περί ασφάλειας, απλά θέλουμε να, καταλάβει, να καταλάβουν οι στρατιωτικές δυνάμεις πώς εμπλέκονται αυτές στη διαδικασία και πώς πρόκειται να εμπλακθούν ενδεχομένως στο μέλλον. Μιλάμε για στρατηγική ανάλυση σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης ώστε να έχουμε καθιδρυμένες διαδικασίες προειδοποίησης και να κατανοούμε που βρισκόμαστε. Αφορά το να κατανοήσουμε, τις, να κατανοήσουμε τη στρατηγική πτυχή των αποστολών. Όταν έχουμε ανθρωπιστική βοήθεια ή βοήθεια μετά από καταστροφή σε διάφορες χώρες που δεν έχουν σήμερα τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν αυτές τις πιέσεις και τις προκλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά ενοποιούνται σε μια στρατηγική σταθερότητα των θαλασσών που υπογράφηκε από τον Υπουργό ε, ε, Εξωτερικών ε, Αμήνης. Πρέπει να φροντίζουμε λοιπόν όλα αυτά να είναι διαθέσιμα στο κατάλληλο χρονικό περιθώριο και να είναι βιώσιμα. Ειδικότερα έτσι εμείς στο στρατό χρησιμοποιούμε την ενέργεια, ο τύπος ενέργειας που χρησιμοποιούμε και η ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιούμε Χρειαζόμαστε να έχουμε τις δυνατότητες και τις υποδομές, αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τη χρησιμοποιούμε με τρόπο βιώσιμο, αποτελεσματικό και χαμηλό, με χαμηλού κόστους για το περιβάλλον. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα. Σημειώνουμε κάποια πρόοδο, όχι σημαντική, αλλά όλο και περισσότερα κράτη συμμετέχουν στο δικό μας σκεπτικό. Θέλουμε τώρα οι άνθρωποι να αρχίσουν να αναλαμβάνουν δράση βάσει αυτού του σκεπτικού και να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία. Εδώ ίσως ε, επισερχείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ στις Βρυξέλλες αλλά και στα κράτη-μέλη. Αυτή η ηγεσία για την οποία ε, μιλήσαμε, να φροντίσουμε, να ε, λειτουργήσουμε ως ομάδα χωρών και να ενθαρρύνουμε τη δράση και σε χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορες δεξαμενές σκέψεις think tanks εργάζονται για αυτό. Δεν είναι αλτρουιστική σκοπή, αφορά και τη δική μας ανάπτυξη, ευημερία και ευεξία. Πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε ωφέλη σε αυτές τις αδύναμες περιοχές και να αξιοποιήσουμε τις συνδέσεις μας, τις σχέσεις μας με την, μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Όπως δείχνει η έκθεση, η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο κοινωνική, οικονομική, υγειονομική, περιβαλλοντική. Υπάρχουν άλλα στρατηγικά ζητήματα σε θέματα ασφαλείας και χρειάζονται δράση για να αντιμετωπιστούν. Όπως δείχνει λοιπόν καταδεικνύει αυτή η έκθεση, οι χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία και άλλες χρειάζεται να κάνουν περισσότερα. Σε ευρύτερο πεδίο, ώστε να ελαττώσουμε τους κινδύνους παγκοσμίους και να αποκομίσουμε τα οικονομικά ωφέλη και την ευημερία που απορρέει από αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, υπονάβαρχε. Ο υπονάβαρχος Μπρούς Βέλχενς αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ίσως θα πρέπει να πω ότι με ενδιαφέρει προσωπικά το θέμα. Είμαι στο ναυτικό, αλλά άρχισα την καριέρα μου ως επιστήμονας οικολόγος και δεν ξέρω που βρίσκομαι τώρα. Είμαστε απολύτως σίγουροι από την οπτική γωνία της ε, στρατιωτικού και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει πάρα πολλά άτομα, όπως και σήμερα το απόγευμα, προηγουμένω δηλαδή, και οι επιπτώσεις για τους στρατιωτικούς είναι πασιφανείς. Αρχίζοντας, θα ήθελα να πω όσο με φορά εμένα κάποια πράγματα γενικά. Το πώς χειριζόμαστε και οι προσδοκίες του πώς χειριζόμαστε εμείς οι στρατιωτικοί της ε, κρίσης που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να σας αφορά και να μπορούμε να διαθέτουμε μέσα εθνικός όταν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Πάντως, όταν δεν μπορούν άλλοι οργανισμοί να προσφέρουν την προστασία από τις επιπτώσεις του κλίματος, τότε είναι σαφές ότι πρέπει να παρεμβαίνει η διεθνής κοινότητα. Και έτσι λοιπόν φτάνω ε, στην ε, δυνατότητα προσαρμογής, ε, την ευελιξία, την οργάνωση όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να επεμβαίνει κανείς με ταχύτητα. Αλλά βεβαίως ε, δεν είναι το απόλυτο για να επιτυγχάνεται η υπόθεση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές ε, του πλανήτη. Ο στρατός λοιπόν ε, θα πρέπει πάντα να είναι σε θέση να ε, συμβάλλει ως ε, ένα είδος ε, διευκόλυνσης στη λήψη αποφάσεων και αυτό μέσα σε μια ευρύτερη προσέγγιση. Τώρα, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την εθνική ασφάλεια, υπάρχουν πολλά καθήκοντα και του στρατού που είναι σημαντικά ή τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Ξεκινώντας λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν τέσσερα στόχοι, τέσσερα καθήκοντα πολύ καθοριστικά ήδη σήμερα για το στρατό που μπορεί να προσφέρει ο στρατός και μπορούν να ε, βελτιώσουν είτε την κοινή ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας είτε τις ε, ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν πληροφορίες που να αφορούν στο περιβάλλον, να υπάρχει σωστή αξιολόγηση του κινδύνου, καθήκοντα που έχουν σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια για να διευκολύνεται η εκένωση του πληθυσμού. Θα αναφερθώ σε όλα αυτά με τη σειρά όπως τα προανέφερα. Ε, πληροφορίες λοιπόν για το περιβάλλον. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει κανείς ε, να συγκεντρώνει πληροφορίες. Η έγκαιρη προειδοποίηση είναι πολύ σημαντική για να γίνεται και η αξιολόγηση κινδύνου. Όσον αφορά τώρα στις ε, περιβαλλοντικές και κλιματικές αλλαγές, οι παρατηρήσεις ε, μας επιτρέπουν να προβλέψουμε τις τάσεις αυτούς τους ε, δύο τομείς. Κατόπιν τούτου, είναι δυνατό να προβλέψουμε καταστροφές. Ο στρατός μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωση αυτή και να εξαλείφουν καλύτερα οι επιπτώσεις από τις περιβαλλοντικές ε, καταστροφές. Ένα πολύ καλό παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της ε, πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει είναι η πρωτοβουλία εκείνη η οποία τελικά ε, θα οδηγήσει στο να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δικές της τις δυνατότητες ε, παρατήρησης γιατί έτσι ε, έχουμε καλύτερη διαχείριση του κλίματος και βελτίωση της ασφάλειας. Επιπλέον αυτή η δυνατότητα οργάνωσης θα επιτρέπει ταχύτερη αντίδραση σε καταστροφές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εξάλλου πέρα από αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη δυνατότητα συνεργασίας. Ε, κατά την άποψή μου μόνο αυτός είναι ο σωστός τρόπος ε, προς τα εμπρός. Και το δεύτερο που θέλω να φέρω έχει την σχέση με την αξιολόγηση των κινδύνων, την ευρύτατη αξιολόγηση. Μία καταστροφή ε, δεν είναι από μόνη ε, σε θέση να μας προστατεύσει από ε, καταστροφές που προκύπτουν λόγω αλλαγών στο περιβάλλον Οι αντιδράσεις θα πρέπει να είναι ενωμένε, να συντονίζονται όλοι οι φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη ή στην άμβλυνση των επιπτώσεων. Να δίδονται απαντήσεις με προστατευτικές δραστηριότητες πρέπει να εντοπιστούν οι δυνατότητες που υπάρχουν, κυρίως όσον αφορά το στρατητικό και δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μοναδική θέση που έχουμε να ε, αντιδρούμε με ταχύτητα σε πιεστικές καταστάσεις ε, Παραδείγματο ε, χάρη ε, να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια και ανακούφιση από τις ε, καταστροφές. Κατά την αρχή των καταστροφών, ο στρατός είναι ο μόνος παράγων που μπορεί να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους έτσι ώστε να υπάρχει ταχεία αντίδραση και βεβαίως έχει και τη δυνατότητα να μετακινηθεί και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως είπα και προηγουμένως. Οφείλουμε βέβαια να αναφέρουμε ότι οι δυνατότητες του στρατού ταιριάζουν και προσφέρονται λόγω της μορφής της οργάνωσης ε, και της ε, φυσικής κατάστασης ε, των ανδρών και γυναικών στο στρατό όσοι πλήττονται από τις ε, καταστροφές ε, κυρίως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Εκεί λοιπόν το να είναι κανείς νέος ίσως να είναι πλεονέκτημα. Οι ε, στρατιωτικές δυνάμεις ε, και η παρέμβασή τους ε, ενδέχεται να μεγαλώσει καθώς ε, θα υπάρχουν όλο και περισσότερες ε, περιβαλλοντικές καταστροφές. Κατόπιν τούτου είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία με τις κυβερνήσεις των κρατών. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα πλεονέκτημα. Ακόμα και αν σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε καταστάσεις που να απαιτούν παραδοσιακές δυνατότητες, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι στο μέλλον ενδέχεται να χρειαστεί κάτι τέτοιο λόγω των αλλαγών, των κλιματικών αλλαγών. Και αυτό απαιτεί και έρχομαι στο τέταρτο σημείο, ε, στο ενδεχόμενο εκένωσης πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών ε, παρεμβάσεων μπορεί να υπάρξει έλλειψη νερού και τροφίμων, ε, είναι σημαντικό να υπάρχει στην αρχή έλεγχος της κατάστασης. Βεβαίως σε τέτοιου είδους περιπτώσεις ε, δεν χρησιμοποιείται ο στρατός για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί αυτό θα υπονόμευε τις προσπάθειες όσων προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Σιγά σιγά όμως, ίσως όπως σας είπα, να κρυθεί απαραίτητο να κενωθούν περιοχές ε, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει το απαραίτητο στρατιωτικό δυναμικό. Και όσον αφορά το δυναμικό αυτό, ε, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το στρατιωτικό δυναμικό. Εξετάζοντας τα διάφορα σενάρια του μέλλοντος, υπάρχει τάση να μιλάει κανείς για την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Ε, οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες που είναι η απόρρια του υπάρχοντος ε, συστήματος και αυτές είναι πάντα σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ε, κλιματικές αλλαγές ε, έγκαιρα. Σε ορισμένα κράτη η κατάσταση ποικίλει, διαφέρει. Έτσι λοιπόν για αυτά τα κράτη ο στρατός είναι ένα, κάτι το πολύ σημαντικό. Παραδείγματος χάρη ενδεικτικά αναφέρω το Μπαγκλαντές οι πληροφορίες για το περιβάλλον και η ευρεία αξιολόγηση των κινητήρων απαιτούν και μία δομημένη προσέγγιση. Ίσως ε, θα πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος οργανισμός ε, υποκείμενος ε, σε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη και το ΝΑΤΟ. Αλλά ακόμα και σε, πρέπει να συμμετέχουν και, και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Η διαμεσολάβηση ε, τρίτων ε, κρατών ε, θα πρέπει να αυξηθεί επίσης έτσι ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε τις συγκρούσεις. Αυτό σημαίνει ότι στις αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπάρχουν και στρατιωτικές γνώσεις. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ο στρατός χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να υποστηρίξει υποβοηθητικά και όχι καθοδηγητικά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, το δυναμικό λοιπόν για τις ε, περιπτώσεις καταστροφής απαιτεί και άλλα πράγματα, όχι μόνο το ε, στρατό, απαιτεί την ανάπτυξη ιατρικών μονάδων και στο τέλος φτάνουμε και στο ενδεχόμενο της εκένωσης. Ίσως ε, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ρεαλιστικές ε, δυνατότητες, να έχουμε τα απαραίτητα σενάρια, μία προσέγγιση που να βασίζεται στην διαπίστωση των αναγκών. Ολοκληρώνοντας λοιπόν θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται τη δημιουργία βάσης δεδομένων ε, που να εντοπίζεται ε, στην ε, επιμελητεία, την υποδομή, στα λιμάνια. Πολύ συχνά, δυστυχώς, δεν είμαστε στο απαιτούμενο επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Κριστιαν Μπρεό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη ευκαιρία για την ΕΑΝΤ που μας καλέσατε να μιλήσουμε για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας στα πλαίσια της ασφάλειας. Θα ήθελα κυρίω να σας πω πώς μπορεί η ΑΕΝΤ να βοηθήσει σε... λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση η οποία γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο λόγια πρώτα απ' όλα για τον τρόπο με τον οποίο οργανούμε. Εμείς είμαστε η υπηρεσία του, Ευρωπαϊκού, του, Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν 26 χώρες πλην της Δανίας. Ε, να κάνουμε ε, έρευνες στον τομέα της δατικής βιομηχανίας, της συνεργασίας και συμφωνούμε απόλυτα με τα οποία, αυτά που προλαεί σα. Αυτέ είναι οι προτεραιότητε του Υπουργού ε, Άμυνα. Προσπαθούμε να κάνουμε συνεργασίε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε με... σε ε, συμμαχικά προγράμματα που αναλαμβάνουμε από κοινού. Προσπαθούμε να αμβλύνουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στη βιοπικιλότητα από την κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις ε, κρίσεις με την ε, ε, μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται και τη μείωση του άχθους το οποίο αφήνουμε με τις δράσεις μας επί τη Η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας έχει μεγάλες επιπτώσεις και στο κόστος. Η ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντική για να φέρουμε σε πέρα στις διάφορες επιχειρήσεις. Η αύξηση της αποδοτικότητας και η μείωση της ε, ε, κατανάλωσης είναι κάτι το πολύ σημαντικό στις περιοχές θεάτρου των επιχειρήσεων και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν προβλέπονται επιθέτης. Επίσης πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τους εξαπλισμούς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Δεδομένου ότι θέλουμε ότι κάνουμε να μην είναι πάρα πολύ βλαβερό για το περιβάλλον. Ποια είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε σωστές λογικές πολιτικές, να είμαστε αποδοτικοί σε θέματα ενεργειακής κατανάλωσης και να δημιουργήσουμε νέα πρότυπα τα οποία θα μας, πρότυπα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε πράσινες λύσεις. Αυτά στα πλαίσια της ε, ευρωπαϊκής ε, πολιτικής που ακολουθούνται και της πολιτικής των μεμονωμένων χωρών. Και σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και θέματα άμυνας υπάρχουν κάποιες ε, αρχές που ακολουθούν όλες οι χώρες. Η θέσπιση πολιτικών και στρατηγικών για τη διαχείριση των κρίσεων σε ευρωπαϊκό κουνδύο μπορεί να είναι ένας σημαντικό κινήτρο για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις βλεπτικές μας, την βλεπτική μας επίδραση επί του πλανήτη μας. Ε, υπάρχουν επίσης ε, πρόγραμμα. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο. Μήπω θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά, σας παρακαλούμε. Κάποια προγράμματα και σχέδια αφορούν επίσης τη γη, τη θάλασσα και τον αέρα. Το θέμα της ε, εξάρτησής μας από τα καύσιμα, ε, εξοπλισμός και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, νέα πρότυπα για την βιομηχανία, είναι κάτι το οποίο ακολουθούμε. Στις 22 Μαρτίου, στα πλαίσια των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άμυνας, τέσσερις χώρες συμμετείχανε στο, έξι χώρες μάλλον, ε, συμμετείχαν στο λανσάρισμα ενός νέου ε, πράσινου σχεδίου. Έτσι, οι στρατιωτικές δυνάμεις των κρατών που έχουν μπορούν βάσει αυτών των σχεδίων που έχουμε να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, συνεργαζόμαστε για την ε, εκπόνηση προγραμμάτων το οποίο ονομάζουμε Military Green 2012. 2020. Στα πλαίσια Επίση, τι ασφάλειες βλέπουμε ποιε είναι οι δυνατότητε που έχουμε για το μέλλον. Αρχίζοντα, θα πρέπει να πω ότι το θέμα των δυνατοτήτων δεν είναι μόνο η τεχνολογία και ο εξοπλισμός. Ο πυρήνα συμπεριλαμβάνει το δόγμα της αντιλήψης, την ετοιμότητα, τη δυνατότητα ανάπτυξης των δυνάμεων και την κατάρτιση όπως είπε και ο κύριος Αμπροζέτη στην αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σχέδιο ανάπτυξη δυνατοτήκη περιέχει, περιέχει μία εκβαθέων ανάλυση του κλίματος στο οποίο εργαζόμαστε και του περιβάλλοντος στο οποίο εργαζόμαστε, λαμβάνει υπόψη διάφορες οικονομικές προβλέψεις, δημογραφικές προβλέψει την ενέργεια, του φυσικού πόρου, το περιβάλλον κτλ. Βάσει λοιπόν των αρχών αυτών έχουν καθοριστεί προτεραιότητες από τα ε, κράτη-μέλη και η, μία από τις ε, δέκα προτεραιότητες τώρα τελευταία ήταν αυτό το θέμα της ε, παροχής ενέργειας, γενικότερα το θέμα των καυσίμων. Τι προσπαθούμε να κάνουμε στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, προβλέψεις, ε, πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, αυτό είναι μία από τι προτεραιότητε που προβλέπει στο τη ανάπτυξή μα. Δεύτερον, πρόληψη και άμβλυνση των φυσικών καταστροφών. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε την επιρροή αυτών των φυσικών ε, καταστροφών και φαινομένων. Τρίτο, αντίδραση σε μια κρίση. Σημαίνει ότι μπορούμε να ε, ηγηθούμε των μέτρων που πρέπει να λάβουμε για να αντιμετωπίσουμε μια καταστροφή. Χρειαζόμαστε λοιπόν δημιουργικό πνεύμα μεταξύ των ε, υπευθύνων και την ανάπτυξη των ε, πρωτοβουλειών από τα ήδη υπάρχοντα όργανα. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε νέες οργανώσεις και όργανα. Τώρα, το θέμα των δυνατοτήτων και των μέσων πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την ε, εκένωση, την παροχή ενέργειας, παροχή ειδών διατροφής και ύδατος, επικοινωνία, ιατρική υποστήριξη, ε, έρευνα, διάσωση, αντιμετώπιση πυρκαγιών, δυνατότητες ανασυγκρότησης και δημιουργίας οδών για την μεταφορά ε, ατόμων και την ε, δημιουργία εκ νέου έργων υπόδομης. Όλα αυτά με τρόπο ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε φυσικές καταστροφές και κατά περίπτωση έναν σεισμό φερρυπίν με τις ιδιαιτερότητες του. Γι' αυτό χρειάζεται και η συνεργασία και οι σαφείς απόψεις της βιομηχανίας. Στην ε, έκθεση ασχολούμαι με το πώς θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει ιδέες το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει και τις δικές μας πτήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα παρόλα αυτά να πω ότι το τι θα γίνει αποφασίζεται από το σύνολο των χωρών που θα μας αναθέσει διάφορα καθήκοντα. Η ΕΑΝΤ θα πρέπει να πω ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μέσο για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του μέλλοντος, κυρίως για να αντιμετωπίσουμε τις, ε, ε, την, τα προβλήματα των κλιματικών αλλαγών, τη βιοπικιλότητα και τα προβλήματα στην ενέργεια. τις ε, υπηρεσίες ε, πυρόσβεσης, ε, ε, έρευνας, διάσωσης, οι ιατρικές υπηρεσίες, ε, υδροδότηση, σύστημα ανείχνευσης για την ε, διάσωση, εκένωση κτλ. Συμπληρωματικά είμαστε το μέσον που μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη δυνατήτων στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής τις βιοπικιλότητες, τις ενέργειες και τις διεθνούς ασφάλειες. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται να υπάρχει βούληση εκ μέρους των κρατών μερών για να μπορέσει η υπηρεσία μας να ενεργήσει και να αναλάβει δερμεύσεις. Το να θεσπίσει πολιτικές και στρατηγικές για την διαχείριση των κρίσεων είναι κάτι που θα μας βοηθήσει να μειώσουμε ε, την αρνητική επίδραση όλων των ενεργειών μας στον πλανήτη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κλερό. Ο κύριος Τόμ Σπένσερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που με να προσδόκηται ο καθεστώς ε, του εμπειρογνώμονα. Δεν είμαι σίγουρος να το αξίζω, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία. Μου κάνει εντύπωση η σημερινή συζήτηση. Αυτή η συζήτηση ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια στη μια συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών και μου κάνει εντύπωση πόσο έχουμε προχωρήσει, προοδεύσει συζητώντας αυτά τα ζητήματα διότι πριν από 10 χρόνια ήταν σαν να βάζουμε μαύρα και ε, άσπρα πετραδάκια πάνω σε ένα πίνακα και να υποθέτουμε πως αυτά θα εξελίσσονταν. Τότε υπήρχε και η έμονη ιδέα με μεγαλύτερη επιρροή του Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και τότε ανησυχούσαμε για τη συμβατότητα των ιδεών μας με τον ΝΑΤΟ. Καθώς ακούω τους συναδέλφους μου μου φαίνεται ότι ασυνείδητα έχουμε δημιουργήσει τους δεσμούς το ε, Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Υπηρεσία Άμυνας, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που τώρα μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε. Όχι να επανειδρύσουμε νέους ε, θεσμούς, να πάρουμε αυτά που έχουμε αντιθέτως και να οικοδομήσουμε επί αυτών. Το Κοινοβούλιο λοιπόν τώρα είναι συνομοθέτης βάσει της Σύνθηκης Λισαβόνας μαζί με το Συμβούλιο. Αυτός είναι ο τρόπος αντιμετώπιση της άμυνας ω θέμα, επειδή η άμυνα πάντα θα χαρακτηρίζει την εθνική ταυτότητα. Η συνεργασία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου μου φαίνεται ότι είναι σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Το ΝΑΤΟ έχει αλλάξει. Ο Τζέισον ίσως από την εμπειρία του στο Αφγανιστάν οι Γερμανοί είναι έτοιμοι να το συζητήσουν στο ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικά ενδεχόμενο στάσει συνεργασία μεταξύ, διάθεση συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς θεσμικών οργάνων, καθώ εξελίσσεται αυτή η ιδέα. Πώ φτάσαμε εδώ. Αρχικά χαρακτήριζε τη δουλειά που ξεκίνησε στι αρχέ αυτού του αιώνα, αλλά και φυσικά με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Περιέργω, μάλλον όχι περίεργος, οι επιπτώσει τη συνθήκη τη Λισαβόνας σε τόσε πολλέ πτυχές επισκιάστηκαν από τη συζήτηση για το ευρώ και την ευρωζώνη, κατανοητό. Αλλά αυτές οι συζητήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν και οριμάζουν. Η έκθεση αυτή θεωρώ περιέχει πολύ κομψά τρία σημεία κλειδιά. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να ε, ευθυγραμμίσουμε, να ομογενοποιήσουμε αυτό το ζήτημα. Να ορίσουμε τις λεπτομέρειες του οικοδομήματος. Υπάρχουν τα διάφορα στοιχεία, τώρα πρέπει να τα συντονίσουμε μεταξύ τους. Και αυτό θα πράξει η Ευρωπαϊκή Πρίση Εξωτερικής Δράσης και όλα αυτά να τα ε, ολοκληρώσουμε με έναν ειδικό εντεταλμένο για το περιβάλλον και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είχα το προνόμιο να παρατηρώ τη δραστηριότητα του πριν τρία χρόνια ε, εξωτερικών υποθέσεων περιβάλλοντος και άμυνας ε, και κοιτώντας το πώς επηρέασε τη διεθνή συζήτηση με, όταν συζητάμε την Αμερική, με τους Κινέζους, με την Νότια Κορέα, με, τους Αυστρα... την Αυστραλία. Είναι εξαιρετικό το να έχει έναν άνθρωπο στον οποίο να μπορούν να εστιαστούν όλα αυτά. Γνωρίζω ότι η δική σα γενιά βουλευτών έχει να αντιμετωπίσει προκλήσει που εμεί δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε τη δεκαετία του 90. Σήμερα πρέπει να ενεργούμε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Ήμουν καθηγητής παγκόσμιας διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Η αλήθεια είναι δεν έχουμε ηγεμόνα, δεν ξέρουμε πώς να λειτουργήσουμε σε ένα πολυπολικό κόσμο και η βασική αιτία δημόσια στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πεποίθηση ότι μπορεί να υπεραμεθεί των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν εξαιρετικά πολύπλοκο κόσμο. Δεύτερον, έχουμε μια τεράστια πίεση να υπερασπίσουμε αυτά που κάνουμε ενώπιον ενός σκεπτικού κοινού, ενός διστακτικού κοινού. Πρέπει τώρα να... Πρέπει να το εξηγήσουμε στην κοινωνία ώστε να ανταποκριθεί η βιομηχανία. Και δεύτερον φοβάμαι ότι η σημερινή γενιά πολιτικών θα έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο 10 χρόνια ύφεση, πολύ χαμηλή ανάπτυξη, αλλά ότι αυτό θα συνεχίσει και στα στη δεκαετία του 2020 όπου θα αρχίσουμε να έχουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να εξοπλίσουμε τους βουλευτές μας και τους υπουργούς μας με επιχειρήματα που να είναι κάτι περισσότερο από ποσοστά. Δεν μπορούμε να προσανατολίζουμε την κοινή γνώμη μιλώντας με ποσοστά. Πρέπει να τους ε, τροφοδοτούμε ισχυρές ιστορίες. Θα σας πω τώρα για ποιο λόγο θεωρώ ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια του στρατού, των στρατιωτικών δυνάμεων. Είναι η μόνη ομάδα που έχει το σεβασμό του κοινού. Εάν πει ο στρατό στην Αμερική ότι οι ανθρώπινε δραστηριότητε προκαλούν κλιματική αλλαγή, το κοινό στην Αμερική θα το πιστέψει παρά την προσπάθεια της βιομηχανίας ε, ορεκτών να τους κάνει να πιστέψουν το αντίθετο. Θέλουμε δηλαδή να δώσουμε δυνατότητες, ενδυνάμωση των στρατών, προπολογισμού. Οι προπολογισμοί αυτοί των στρατών είναι τεράστιοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ε, υποδομών αποθήκευσης ας πούμε ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια. Τρίτον, θέλουμε το στρατό ως υπόδειγμα εάν ο στρατός μπορεί να μεταρρυθμιστεί, να ελαττώσει τις ανθρακούχες εκπομπές, να μειώσει τον προϋπολογισμό ε, εγκαταλείποντας τα ορεικτά καύσιμα, αυτό θα επηρεάσει όλους και θα ενθαρρύνει όλους. Δηλώνουμε αυτά που ξέρουμε για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την αποτυχία των κρατών, οδηγεί τους ανθρώπους στη μετανάστευση. Κατά την άποψή μου, και χαίρομαι που αναφέρεται στην έκθεση, δεν είναι απλά πολλαπλασιαστή των απειλών. Μπορεί να αποτελέσει κρίση από μόνο του. Στις ε, αρχικές αναφορές σε κλιματικές αλλαγές, στις αρχικές εκθέσεις, αναφερόταν ως απειλή. Σήμερα είναι πολύ περισσότερο από, μια, από πολλαπλασιαστής απειλής. Έχω να σας πω μια ιστορία από την Ασία για να δούμε τις πραγματικές διενέξεις σειράξεις για τα επόμενα 40 χρόνια θα χρειαστεί να στραφούμε στην αστάθεια που θα παρατηρηθεί στη Δυτική Κίνα, στην Αγροτική Ινδία λόγω της αδυναμίας παροχής νερού. Ποια θα είναι η κινέζικη απάντηση θα ανοίξει μια τρύπα στα Ιμαλάια και θα αλλάξει ε, το ρου του Βραχμαπούτρα. Εάν γίνει αυτό μπορώ να σας πω ποια μονάδα τη Ινδικής αεροπορίας θα βομβαρδίσει αυτό το φράγμα. Εάν ε, τραβήξουμε τα νερά αυτά μακριά από τον Μπαγκλαντές ε, θα μπορούν να περάσουν εκατομμύρια ε, κατοίκων του Μπαγκλαντές από τα σύνορα τι πρέπει να κάνουν οι Ινδοί σε αυτή την περίπτωση, τι πρέπει να κάνουν οι Κινέζοι εάν η σταθερότητα στη Δυτική Κίνα διαταραχθεί. Αυτά είναι τεράστια ζητήματα και θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Εγώ είχα ασχοληθεί με όλο αυτό στο αντίστοιχο συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε. Έχω σχεδόν εξαντλήσει το χρόνο μου. Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι όταν λέμε μια ιστορία στους Ευρωπαίους πολίτες πρέπει να δείχνουμε πώς επηρεάζονται οι Ευρωπαίοι σήμερα. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι απόμεκρο που συμβαίνει μόνο σε αναπτυσσόμενες χώρες. Μπορεί να μας επηρεάσει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που θα βρει μεγάλη απίχυση στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή εξαρτόμαστε για τους σωλήνες μεταφορά φυσικού αερίου για την παροχή του φυσικού αερίου. Αυτοί βρίσκονται πάνω στο πέρμαφρος, καθώς το πέρμαφρος θα, λιώνει, θα λιώσει, θα διακοπούν αυτοί οι σωλούνες. Συνεπώς αυτή η προφανής μας ασφάλεια είναι απατηλή. θα υποφέρουμε από τις κλιματικές αλλαγές, θα υπάρξουμε θύματα και αυτό θα φανεί και με την έκθεση αυτή έχουμε την ευκαιρία να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά και να τα εκφράσουμε με έναν τρόπο που θα τον κατανοήσουν οι πολίτες της Ευρώπης. much, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σπένσερ. Ακούσαμε λοιπόν ε, τέσσερις ε, ολοκληρωμένες εκθέσεις με πάρα πολλές και συγκεκριμένες ε, απόψεις και πολλές νέες ιδέες. Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι θα έχουν να υποβάλουν ερωτήσεις, αλλά αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε αργότερα. Τώρα λοιπόν ε, προτείνω να λάβουν το λόγο οι σκιώδεις εισηγητές επί του, επί του θέματος που συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις σας σε αυτή την συνεδρία των εμπειρογνωμόνων για τις πολύ πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Γιατί όλες αυτές οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν στο να καταθέσουμε τις τροπολογίες μας στην έκθεση. Και θέλω λοιπόν εδώ να σας κάνω και κάποιες επιπρόσθετες ερωτήσεις ε, και θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω τα σχόλιά σας. Καταρχήν, στην πρακτική, πώς ακριβώς βλέπετε τη συνεργασία ανάμεσα στις ε, στρατιωτικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τις πολιτικές μονάδες όπως είναι η Γενική Διεύθυνση ε, περι Περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συνεργασία και να μην υπάρχει και επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Δεύτερον, η επόμενη ερώτησή μου είναι λοιπόν η εξής. Εάν η εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας δραστηριοποιηθεί περισσότερο στην περίπτωση των περιβαλλοντικών καταστροφών, πώς μπορούμε και να διασφαλίσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές ε, οι στρατιωτικές δυνάμεις αντί να βοηθήσουν παρεμποδίζουν το έργο των υπολείπων. Ίσως ε, αυτή η ιδέα της ε, ε, παροχής στρατιωτικής βοήθειας ε, για περιβαλλοντικές καταστροφές να αντιβαίνει σε άλλες βασικές αρχές. Στην έκθεση γίνεται και για την αποστολή εμπειρογνωμόνων, αλλά ίσως θα ήταν πιο αποτελεσματικό εάν προετοιμάζαμε το προσωπικό μας, τις αντιπροσωπείς που στέλνουμε, να αναλύουν την κλιματική αλλαγή για από το πρίσμα της ασφάλειας, έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα των καταστροφών, αντί να προκαλούν περισσότερη γραφειοκρατία. Στη τελική ανάλυση ε, ε, είναι απαραίτητο να υπάρχει μία εμπεριστατωμένη μελέτη και θέλω να υπογραμμίσω ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε καλύτερη πρόληψη, διότι αυτό είναι πολύ πιο φτηνό από το να αντιδρούμε ad hoc σε φυσικές καταστροφές. Εδώ λοιπόν επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι ε, η ε, ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας δεν έχει άμεση σχέση με την πρόληψη. Σε ευχαριστώ κύριος Βότσον. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ προς το παρόν. Η κυρία Λέζινγκ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι και πάλι ε, πολυεπίπεδο. Ε, βεβαίως ε, πρόκειται εδώ για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για την πρόληψη. Ίσως εδώ να μην είναι η κατάλληλη επιτροπή για να συζητήσουμε το θέμα, παρότι είναι το θέμα σημαντικό. Για μας λοιπόν τι ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι το αστικό, το πολιτικό σχέλος, ποιο είναι το στρατιωτικό, τι είναι η οικολογική καταστροφή, γιατί πολλές φορές ε, αναφέρεται ότι ο στρατός έχει το καλύτερο δυναμικό για να βοηθήσει. Κατόπιν τούτου, για να υπάρχει αποτελεσματική παροχή βοήθειας, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται οι στρατιωτικές δυνάμεις. Αναφέρθηκε ότι είναι σημαντικό να ε, εντάξουμε διάφορα και διαφορετικά στοιχεία κάτω από μια συγκεκριμένη ομπρέλα. Αυτή η ομπρέλα θα πρέπει όμως ε, να παρεμβαίνει σε καταστροφές ε, και όχι να διοχετεύουμε όλο και περισσότερα κονδύλια σε στρατιωτικές δυνάμεις, έτσι ώστε τελικά να παρεμβαίνουν οι πολιτικές. Κατά την άποψή μας, αυτό είναι κάτι θεμελιώδες. Κάτι άλλο που θέλω να φέρω είναι το εξής. Από όλα αυτά τα σενάρια που ακούσαμε, ποιο είναι το πραγματικά στρατιωτικό. Αναφέρθηκαν λέξεις κλειδί, όπως ε, η περίφημη λέξη κλειδί «καζούς μπέλι». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Εάν κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, ας δούμε λιγάκι αυτό το χάρτη. Ε, εφόσον τίθενται σε κίνδυνο εμπορικές οδοί, τι σημαίνει αυτό κάτω από ε, στρατιωτικό πρίσμα. Τι σημαίνει ότι μπορούν να υπάρξουν εδαφικές απώλειες. Αυτές δηλαδή οι εδαφικές απώλειες θα προκύπτουν ή θα εξισορροπούνται με στρατιωτικές παρεμβάσεις. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο. Ε, πρέπει να το συζητήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι την άποψή μας από αυτού του θέματος ε, τη γνωρίζετε. Εδώ ως ε, πανάκια αναφέρεται το περίφημο pooling and sharing. Κατά τη δική μας άποψη αυτό το pooling and sharing αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και την κατανομή των εξουσιών που, εν πάση περιπτώσει, είναι και ο πυλώνας της δημοκρατίας. Θα ήθελα να τρέξω ε, και σε ένα παράδειγμα από το παρελθόν. Στην Αιτή συγκεκριμένα. Εκεί στην Αιτή τι ρόλο έπαιξε ο στρατιωτικός. Πώς προστάτευσε από την καταστροφή. Γιατί είχαμε πλοία ε, μπροστά από, στο λιμάνι της ε, ΑΕΤ που φιλοξένησαν προσφύγους. αυτό το σκέλος νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμο. Εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στρατιωτικό στοιχείο για, στην περίπτωση οικολογικών καταστροφών. Οι ε, στρατιωτικές δυνάμεις ε, που έχουν και ιατρική υποστήριξη θα μπορούσαν ίσως να περιθάλψουν τραυματίες, επειδή όμως δεν υπήρχαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν προσέφεραν βοηθείς. Εγώ τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ε, μέσω των ε, φυσικών καταστροφών υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιούνται στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες όμως προσχηματικά τα χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους καταστροφές. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην ανακατεύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις με την ε, αστική πολιτική ε, παρέμβαση και να μην υπάρχουν και συγκαλυμμένοι ε, προπολογισμοί εξοπλισμών. Αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω στον εισηγητή. Αυτό το θέμα του ταμείου που έδειξε, πώς ακριβώς το σκέφτεται. Αυτό το ταμείο, τι θα χρηματοδοτεί. Και οι γραμμές αυτές του προϋπολογισμού, ε, πώς θα διαμορφώνονται, πώς θα πρικοδοτούνται. Είμαι και εγώ σκιώδης εισηγητής για την έκθεση αυτή εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Και μπόρεσα να εκφράσω απόψε τον κύριο Τάνταν, πλήρως υποστήριζε την έκθεσή του και νομίζω ότι όση προσοχή και να δώσουμε στην κλιματική αλλαγή, ποτέ δεν ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε αρκετά. Το πρόβλημα μας το μεγάλο τώρα είναι η οικονομική κρίση. Για να εξοικονομήσουμε χρόνο στη σύστη θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να κάνουν σχόλια για την έκθεση, για τις και παρατηρήσεις σύντομα και κυρίως να κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τους ε, τέσσερις εμπειρογνώμονες οι οποίοι μας ε, παρουσίασαν την πραγματική διάσταση του θέματος και οι ε, οποίοι, οι επίσης μας έδειξαν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πολιτική. Θα ήθελα, σε σχέση με αυτά που λέξαμε προηγουμένως, να πω το εξή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της Ένωσης υπάρχουν δύο βασικές αρχές. Η μία αρχή είναι ότι υπερισχύει η πολιτική. Δηλαδή, δεν ισχύει αυτό που ισχύει σε άλλες χώρες ότι υπερισχύουν οι στρατιωτικοί και υποτάσσονται οι πολιτικοί. Η υπεροχή της πολιτικής σημαίνει ότι το στρατιωτικό, οι στρατιωτικές δυνάμεις υπάγονται απόλυτα στους ερετούς εκπροσώπους των πολιτών. Σε εμά λοιπόν, οπουδήποτε χρησιμοποιούνται στρατιωτικές δυνάμεις, αυτό γίνεται μετά από απόφαση της, ε, νομικά, της ε, νομιμοποιημένης πολιτικής ηγεσία, όχι αντίστροφα. Και κατόπιν υπάρχει και η αρχή της διαφάνειας του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι τόσο ο προϋπολογισμός εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και αυτή των ε, κρατών μελών χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, ε, λογοδοτούν οι αρμόδιοι στις ε, κυβερνήσεις, ε, στα κοινοβούλια. Πάντως ε, και αυτό είναι ένα στοιχείο, υπάρχουν εχέγγυα, ότι αυτά δηλαδή που διαδραματίζονται σε στρατιωτικό τομέα είναι η έκφραση της πολιτικής βούλησης. Όχι δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην Αίγυπτο, στη Πακιστάνη, οπουδήποτε αλλού, όπου ε, ισχύει το αντίθετο. Εμείς δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Γι' αυτό λοιπόν, κατά την άποψή μου, είναι σωστό, απαντώντας την ερώτηση του πώς θα αντιδράσουμε ε, σε αυτές τις ε, προκλήσεις, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε σωστά τα εργαλεία μας είτε πρόκειται ε, για μία πλημμύρα ε, στην ε, Πολωνία, είτε πρόκειται για υπερχείληση ποταμού στη Γερμανία, είτε έρχονται οι διασώστες από τη Γερμανία, είτε είναι στρατιώτες, είτε αστυνομία. Ανεξάρτητα με όλα αυτά πρέπει να υπάρχει η πρόσκληση και η πολιτική βούληση εκείνων που προσκαλούν τις δυνάμεις. Αυτό δεν το βρίσκω κακό ή αντίστροφα αν το πάρετε σε τρίτες ε, χώρες ε, ξεσπάνε ε, πυρκαγιές οι οποίες οδηγούν σε μαζικές μετακινήσεις προσφύγων. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν σήμερα εργαλεία με βάση τα οποία είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε και να αντιδράσουμε. Είναι αδιάφορο το κατά πόσον το αίτιο είναι φυσική καταστροφή που προέρχεται από κλιματική αλλαγή και ξεσπάει φωτιά ή αν υπάρχει ένας εμπριστής ε, που βάζει φωτιά ε, σε τελική ανάλυση είναι ένα και το αυτό γιατί τα εργαλεία που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις δύο περιπτώσεις είναι ακριβώς τα ίδια. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δίνουμε τις απαντήσεις ε, με βάση τις δυνατότητες μας. Στην προηγούμενη συζήτηση που προηγήθηκε ε, έγινε λόγος για το GMS, ε, συζητήθηκε το κατά πόσον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αυτό στον προϋπολογισμό μας, να δούμε κατά πόσον εμείς ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε εργαλεία τα οποία να μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά όλες αυτές τις ε, προκλήσεις. Όσον αφορά την έκθεση Τάραντ, η εισηγήτριά μας, κυρία Νάνσκι, νομίζω ότι τοποθετήθηκε από αυτού και γνωρίζω ότι έχει προετοιμάσει μια σειρά πολύ καλών τροπολογιών που θα καταθέσει έγκαιρα. Εμείς λοιπόν ως ε, ΕΛΚ θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Στάνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η πρώτη φορά που διαβάζω την έκθεση Τάντρα και είναι συναρπαστική. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω τρεις συμπατριώτες μου εδώ από το Ηνωμένο Βασίλειο και που μας μιλούν για αυτό. Τον κύριο Μορσέτη είχα την τιμή να τον γνωρίσω πέρυσι, έτσι γνώριζα ήδη τη θέση του και το μακροπρόθεσμο σκεπτικό σε αυτό το τομέα. Η ερώτησή μου προς αυτόν είναι το Υπουργείο Αμήνης του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή η θέση που ε, εφαρμόζεται και σε άλλα Υπουργεία Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Υπάρχει περίπτωση επικάλυψης μεταξύ του ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκής ένωσης η Συντονίζεται όλο αυτό το σκεπτικό μεταξύ των δύο ε, στρατιωτικών συμμαχιών. Σε ποιο βαθμό όχι συμμαχία, λάθος λέξη, το ΝΑΤΟ είναι συμμαχία ουσιαστικά, αλλά τα προγράμματα κοινή άμυλα και ασφάλεια ε, είναι μια πολιτική ουσιαστικά το CSDP ε, πρόγραμμα το οποίο να περιλαμβάνει στοιχεία που το κάνουν να λειτουργεί σαν συμμαχία ορισμένες φορές. Ε, αυτό με ενδιαφέρει διότι Συμπτωματικά αυτή την εβδομάδα έχω την εκθεσή μου για το ε, Βόρειο Αφρική, για το κέρας της Αφρικής. Δεν έχω αναφέρει αυτό το ζήτημα καθόλου στο σχέδιο εκθεσή μου και παρατηρώ εδώ στην παράγραφο 5 μιλάει για το κέρας της Αφρικής συγκεκριμένα. Ίσως αυτό θα ήταν κάτι που καλό θα ήταν να συμπεριλάβω δεδομένη του στρατηγικού χαρακτήρα της περιοχής με την Ερθρά Θάλασσα, το κανάλι του Σουέζ, τους θαλάσσιους διαδρόμους και το τι έρχεται από νότια όσον αφορά το πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο και τον Αραβικό κόλπο. Τι σημαίνει αυτό με τις μαζικές μεταναστεύσεις ανθρώπων λόγω λοιμού ή άλλων αλλαγών ή σειράξεων στην περιοχή. Εγώ είμαι τη σχολή ε, όπως σκεπτόμαστε ότι ίσω δεν μπορούμε να κάνουμε και τόσο πολλά για να σταματήσουμε την ε, υπερθέρμανση του παλίτη, ο μετριασμός δεν είναι πολύ εύκολος σε περίπτωση που τα χειρότερα σενάρια γίνουν πραγματικότητα όποιες και είναι οι απόψεις σας για το κατά πόσο είναι ανθρωπογενές αυτό ή όχι ή κατά πόσο προέρχεται από τον ήλιο μου φαίνεται ότι θα είναι οικονομικά εξαιρετικά δύσκολο να καταπολεμηθεί επαρκώς. Θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη λαμβάνει τη δέσμευση των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω το ITER που είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο θεωρώ ότι προληπτικά πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα πράγματα και τι πρέπει να γίνει όχι να σταματήσουμε φυσικά την κλιματική αλλαγή αλλά πώ μπορούμε να λάβουμε μέτρα ασφαλεία και άμυνα ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα σενάρια και να διασφαλίσουμε τα οικονομικά και εμπορικά μας και λοιπά συμφέροντα. Αυτό μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον και ένα σας ρωτάω τι κάνει το ΝΑΤΟ, τι κάνει η CSDP, ε, τι γίνεται με τη CSDP στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάμπελ Μπάνερμαν παρακαλώ. Με, ναι, κύριος Κάμπελ Μπάνερμαν, συγγνώμη, ζητάει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φοβάμαι ότι εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη. Θεωρώ ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ήμουν μόλις τόσο σε τον Βίκινγκ στη Δανία, όπου η, κλιματική αλλαγή για αυτούς ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν όταν η Γρυλανδία πρασίνησε και ε, εμείς ε, έχω τεράστιο σεβασμό προς ε, τους ομιλητές μας εδώ Αυτό που με ενδιαφέρει γνωρίζουμε ότι θα γίνουν αυτά, θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Λοιμούς, σεισμοί, τσουνάμι. Σίγουρα καλό θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους ε, διεθνή δύναμη διάσωσης ε, μια διεθνής δύναμη που θα μπορεί να δραστηριοποιείται πολύ γρήγορα με ελικόπτερα έτοιμα, με θαλάσσια μέσα, νερό, τροφή, καταλήματα. Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά θα συμβούν, οτιδήποτε και αν τα καθοδηγεί αυτά, είτε πρόκειται για την κλιματική αλλαγή είτε για κάτι άλλο. Είμαι βέβαιος ότι μιλάμε εδώ πέρα για μια διεθνή δύναμη στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Υπάρχει λοιπόν κάποιος προβληματισμός για... προς αυτή την κατεύθυνση, διότι έχουμε ακούσει πολλά αλλά μπορούμε, υπάρχει δυνατότητα ταχείας απόκρισης εντός αεροδοκτορών ε, ε, και η στρατιωτική είναι, η στρατό είναι ουσιαστικά ο μόνο που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Λέζινγκ, παρακαλώ ξανά. Ναι, Κοιτάξτε, ε, θα ήθελα να πω στον κύριο Τένοκ ότι του είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που μου είπε. διόρθωσε αυτά που είπε. Κοιτάξτε, ως ψυχίατρος ε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ε, και αυτό που υπάρχει το φροηδικό λάθος ε, Θεωρώ λοιπόν ότι και το φροηδικό λάθος έχει και αυτό κάποια αξία. Μία ερώτηση προς τον κύριο Γκάλα. Είπατε προηγουμένως ότι Οτιδήποτε άπτεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύεται από διαφάνεια. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άλλα κράτη όπου η κατάσταση είναι χειρότερη. Αλλά ξεχάσατε τι συζητάγαμε εδώ σήμερα το πρωί. Αυτό ακριβώς το ε, θέμα ήταν το πρόβλημα. Ότι δηλαδή στις γραμμές του προπολογισμού δεν αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια ποιε είναι, ποιες είναι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ποιες είναι πολιτικές. Και κάτι άλλο. Ε, όσον αφορά το περίφημο pooling and sharing. Κοιτάξτε, όλο το, σύνολο του δυναμικού μπαίνει σε μία δεξαμενή και μετά κατά κάποιον τρόπο αποφασίζεται το ποιο θα πάει πού. Πώς είναι δυνατόν εκεί να υπάρχει διαφάνεια. Ίσως μπορείτε λιγάκι να μου το εξηγήσετε. Ίσως εγώ να κάνω λάθος. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο ε, που το ξέχασα προηγουμένως, οι εμπειρογνώμονές μας είπαν ότι στην κοινωνία και υποθέτω ότι εννοούν την ε, κοινωνία των ε, πολιτών. Ε, η κοινωνία των πολιτών κτιμά ιδιαίτερα την παρέμβαση στρατιωτικών και ότι οποτεδήποτε κρίνεται αυτή απαραίτητη την αποδέχονται. Αυτό όμως εγώ το αμφισβητώ γιατί πρέπει να σας πω ότι αν γίνουν έρευνες θα προκύψει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Και στη Γερμανία συγκεκριμένα το 80% ε, όταν, ε, όσων ερωτήθηκαν είπαν ότι ακριβώς στο στρατιωτικό τομέα επιθυμούν να υπάρξει εξοικονόμηση κονδυλίων και επιθυμούν τα κονδύλια να χρησιμοποιούνται σε άλλους τομείς και μετά αναφέρθηκε ότι απλά πρέπει κανείς να το εξηγήσει στους ανθρώπους. Αυτό όμω είναι μεγάλος κινδύνος να δούμε που ακριβώς υπάρχουν σημαντικοί στόχοι και μετά ε, να λέμε ορισμένα πράγματα σε ανθρώπους που ούτε καν να ισχύουν. Γι' αυτό λοιπόν ε, υποβάλλω εκ νέου την έκκληση να υπάρχει ως το δυνατόν ε, μεγαλύτερη ασφάλεια. Διαφάνεια, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, καταρχήν, όσον αφορά στον προϋπολογισμό, ε, στην ε, εκτέλεση του προϋπολογισμού έχουμε τη δυνατότητα εμείς ε, ως ε, κοινοβούλιο να ε, μπορούμε να ελέγχουμε τα πράγματα. Εκεί λοιπόν έχει βελτιωθεί η κατάστασή μας και εκ των υστέρων υπάρχει ο δημοσιονομικός έλεγχος και οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ αυστηρές. Το πρόβλημα είναι ότι ε, δεν διοχετεύονται κονδύλια διότι οι διαδικασίες είναι τόσο περίπλοκες που τελικά δεν φτάνουμε στο να εκταμιεύονται τα κονδύλια. Εγώ λοιπόν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Πράγματι μπορούμε να παρακολουθήσουμε ε, το τι ακριβώς ε, φεύγει από τον προπολογισμό μας. Ε, το pooling και sharing αυτά είναι πράγματα που λαμβάνονται, λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του προπολογισμού στους εθνικούς προϋπολογισμούς και μετά υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα όπου συμφωνούν περισσότερα κράτη-μέλη είτε να συγκεντρώσουν τις ε, δυνάμεις τους έτσι ώστε να έχουν ε, ένα, μια ισχυρή, ένα ισχυρό δυναμικό ή υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι κοίταξε θα σε βοηθήσω. Ε, το ΝΑΤΟ παραδείγματος χάρη είναι μια πολύ καλή ένα πολύ καλό παράδειγμα, οι αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Αντί να αρχίσει τώρα η Λιθουανία και η Λετωνία να έχουν τη δική τους στις δικές τους αεροπορικές δυνάμεις, καλύτερα να το αναλαμβάνουν κάποιοι άλλοι και να εξασφαλίζουν την ε, ε, ασφάλεια. Το pooling and sharing θέλουμε επιτέλους να ελπίζουμε ότι θα προκαλέσει την απαραίτητη εμπιστοσύνη, γιατί εδώ και 70 περίπου χρόνια έχουμε ε, ειρήνη και έτσι λοιπόν ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, ακόμα και αν κάποιο το επιθυμούσε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον ε, ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν, Γενικό Διευθυντή της ΕΚΟ, επικεφαλής τον κύριο Χαβιέ Πέρες Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω επί τη ευκαιρία τον κύριο Ταράντ που μας εισάκουσε όπως ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του. Όπως είπε ο κύριος Ταράντ, ήρθε σε επαφή με τις ε, πολιτικές υπηρεσίες της Κομισιόν και σίγουρα με τους συναδέλφους ε, από την Διευθύνση Κλιματικής Αλλαγής ότι άκουσε ότι χαίρονται που η έκθεση αυτή θέτει επιτάπητος ε, αυτό το παγκόσμιο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ειρήνη και στη σταθερότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, θα θέλαμε να τονίσουμε, όπως είπαν και άλλοι συνομιλητές νωρίτερα, ότι έχουμε πολλά χρόνια εμπειρίας στο διεθνές προσκήνιο όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Θα θυμάστε το 2010 δημοσίευσε μια ανακοίνωση η Κομισιόν για την ε, αύξηση της αποτελεσματικότητας της ε, αρρωγής σε περίπτωση καταστροφών και της απόκρισης σε καταστροφές και επανεξετάζουμε τώρα το μηχανισμό στο Κοινοβούλιο. Ε, όλα αυτά είναι μέσα που θα θέλαμε να θέσουμε σε συζήτηση ώστε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση καταστροφών. Θα θέλαμε επίσης ε, να τονίσουμε το ρόλο της ε, Κομισιόν ε, τα τελευταία χρόνια ε, για την απόκριση σε φυσικές καταστροφές μέσω των δύο μέσων που χρησιμοποιούμε την πολιτική προστασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. Τέλος, στο σημερινό διεθνές πλαίσιο σύστημα ουσιαστικά αυτής της απόκρισης σε περίπτωση καταστροφών θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η χρήση στρατιωτικών μέσων διεθνών στρατιωτικών μέσων για ρογή σε περίπτωση φυσικών καταστροφών σε διεθνές επίπεδο όπως ανέφεραν ορισμένοι συνάδελφοι καθοδηγείται από διεθνείς κατευθύντηριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν και αυτό το ανάγκη σεβασμού τήρηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Όπω είπαν οι συναδέλφοι από τα στρατιωτικά επιτελεία, ο κ. Βίλιαμ. και πιστεύω πολύ σωστά η στρατιωτική ο στρατός θα υποστηρίξει, δεν θα ε, ηγείται της απόκρισης ε, σε περίπτωση ανάγκης ε, ανθρωπιστικής αρρωγής. Η απόκριση σε περίπτωση καταστροφών. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η κυρία Εύα Κόρδοβα, παρακαλώ. Ε, good afternoon. Γεια σας, θα πω, θα πω δύο-τρία γενικά σχόλια πριν να δώσω το λόγο στον συνάδελφο που ασχολείται με την κλιματική αλλαγή. Απλώς θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζουμε το ότι συζητείτε αυτό το θέμα εδώ για ε, την άποψή μας θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο με στο οποίο θα χειριστούμε όλα αυτά τα σημαντικά θέματα. Και αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι, όπως λέγεται και στην έκθεση, ε, διεξοδικό και συνολικό. Για την επίλυση της κρίσης στην Ευρώπη έχουμε τους διάφορους φορείς οι οποίοι θα πρέπει να συνεισφέρουν, να εμπλακούν στις δράσεις, όχι σε ιστορικό επίπεδο, αλλά σε εξωτερικό δεδομένο ότι μιλούμε εδώ για την εξωτερική διάσταση του όλου θέματος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε με τον κατάλληλο τρόπο στην διαχείριση αυτή της κρίσεως, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, οι σωστοί άνθρωποι να είναι σωστές θέσεις και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε περαιτέρω να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που πραγματεύεται η έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτιν Φέλτς. Γεια σας, θα ήθελα να πω ότι ήδη έγινε πέρσι στο Συμβούλιο Εκτορικών επαθέσεων. συζήτηση το θέμα αυτό της ασφάλειας που μπορεί να προέρχεται από κλιματική αλλαγή και για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα, τρεις διαφορετικές δράσεις θα πρέπει να αναλυφθούν. τρεις άξονες διαφορετικοί. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, που έχει δυνατότητες να μπορέσει να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αυτών που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις για να σιγουρευτούμε ότι αυτοί οι οποίοι ξέρουν και λαμβάνουν αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις ξέρουν περί τίνος πρόκειται και να γίνουν διάφορες ε, ε, σημαντικές προσαρμοτικές ε, προσαρμογές. Όλα αυτά της κλιματικής, αν θέλετε, διπλωματίας είναι θέματα με τα οποία ασχολεί το Συμβούλιο των Υποθέσεων έχει αρχίσει πολιτικός διάλογος με κάποιες χώρες στις ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται ευρύτατα και είναι και θέμα της ε, συνεργασίας την οποία έχουμε με διάφορες ε, άλλες τρίτες χώρες του κόσμου και υπήρους όπως χώρες κεντρικής ε, Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτή την σφαιρική προσέγγιση και να δημιουργήσουμε κίνητρα ώστε συλλογικά όλο και περισσότεροι γιατί να ασχοληθούν διεθνώς με το θέμα αυτό της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Υπάρχουν κάποιες ιδέες και συστάσεις στην έκθεση που θα εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή. Ένα μέρος αυτών είναι θέμα και συντονισμού της ΕΑΤΣ μεταξύ κρατών μελών. Λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα οποία λέγονται και πρέπει να πω ότι είναι και μέρος των εργασιών με τις οποίες εμείς ασχολούμαστε. Πριν να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, θα ήθελα και εγώ να κάνω μία ερώτηση. Έξι ή επτά χρόνια πριν, ο κύριος Χαβιέρ Σολάνα είπε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ασφάλεια είναι η κλιματική αλλαγή. Αυτό ισχύει τώρα, ισχύει περισσότερο, ισχύει λιγότερο. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε μπροστά αυτή την κατάσταση. Κύριε Μωρισέτη, έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλια που έγιναν. Ήταν απλά τα πράγματα όταν πήγα εγώ στην αρχή στο ναυτικό. Είμαστε μια στρατιωτική συμμαχία 12 κρατών και το βασιλικό ναυτικό είχε πολύ λίγα προβλήματα. Μετά έγιναν ε, τα πράγματα πιο πολύπλοκα, συνεργαστήκαμε με την αεροπορία, προχωρήσαμε σε νέες συμμαχίες. Σήμερα έχουμε άλλες κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές συμμαχίες και ενεργούμε σε πολύ περισσότερους άξονες. Αυτές είναι μεγάλες προκλήσεις. Εδώ δεν μιλούμε για συμπληρωματικούς πόρους για το στρατιωτικό τομέα. Θέλουμε με τα υπάρχοντα μέσα που έχουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο που μπορεί να απορρέει από την κλιματική αλλαγή και να βοηθήσουμε και την ε, οικονομική ε, κατάσταση. Ε, κοιτάξτε, οι στρατιωτικοί μπορούν να βοηθήσουν. Κοιτάξτε με την ηγεσία των, των πολιτικών πόσο καλά βοήθεια μπορούμε να, πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε στην παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και εδώ μπορούμε λοιπόν κάτι να κάνουμε. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποια είναι και οι κίνδυνοι σε περιοχές που έχουμε ε, δυνατότητα ανάπτυξη σειράξεων. Και εκεί θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη συνεργασία. Και θα σας ε, αναφέρω το θέμα το οποίο δημιουργείται στην, ε, στο κέρας της Αφρικής, στην γειτονική Σομαλία, στα προβλήματα στα οποία δημιουργούνται και στο πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Με άλλους φορείς και οι ε, στρατιωτικοί μπορούν να βοηθήσουν στο να είναι ε, καθαρά τα ύδατα, να είναι πόσιμο το είδος, να βοηθηθούν η ε, τοπική παραγωγή, αλληλείς, γεωργοί Πρόκειται για μια περιοχή η οποία πλήττεται πάρα πολύ από την κλιματική αλλαγή. Όχι μόνο διότι προκαλεί στις χώρες αυτής της Κεντρικής Αφρικής ε, τρομερά ε, προβλήματα όσον αφορά τα είδη ε, διατροφής, αλλά διότι μπορεί να αποτελέσει γενικότερο κίνδυνο για όλη την περιοχή. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό τι είδου μηνύματα θα στείλουμε και σε αυτέ τι χώρε. Και κυρίω τι μηνύματα θα στείλει η ΕΠΑ για θέματα ασφαλεία. Θα πρέπει να σταλούν τα σωστά μηνύματα με τη σωστή γλώσσα για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτούς τους λαούς. Τώρα, να αφαιρθώ σε κάτι πιο ειδικό. Αυτό το οποίο ελέγχθη προηγουμένως για τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών για τις Green Barriers είναι ε, ένα σημαντικό θέμα. Ξέρουμε ότι με αυτά τα θέματα ασχολούνται και διάφορες περιφερειακές δυνάμεις. Θα πρέπει όμως αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε δράσεις που να βοηθήσουν πραγματικά τους λαούς οι οποίοι πλήττονται από όλα αυτά τα προβλήματα. Και εδώ μπορεί κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσει δευτερευόντως και ο στρατός. My role around the world Πρέπει να πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μοναδική χώρα που έχει κατά κάποιο τρόπο έναν ειδικό απεσταλμένο για τέτοιου είδους ε, θέματα για να αντιμετωπίσει ε, αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και εκ μέρου του στρατού και εκ μέρου του ναυτικού υπάρχει κάποιο που ασχολείται με αυτό το θέμα. Πολλοί ασχολούνται λοιπόν με το θέμα αλλά μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωση νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα πραγματικής συνεργασίας για να αντιμετωπιστούν όλες οι προκλήσεις και για να εξασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους που διαθέτουμε. Συμπεραίνοντας, θα πω ότι φαίνεται στην έκθεση ε, ότι αναφέρονται τα πιο κύρια θέματα στα οποία πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Πολλά θέματα καλύπτονται στην έκθεση και νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. So, uh, Admiral, uh, Bruce Williams. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις θα ξεκινήσω με κάποια σημαντικά σημεία που ανέφερε η κυρία Λέζιν. Μου έκανε εντύπωση η σκέψη σε σχέση με το μέγεθος ε, του στρατού και τον πόρο του στρατού. Αντιλαμβάνομαι ότι ε, ο στρατός σήμερα είναι κλάσμα του στρατού που ήταν όταν εγώ μπήκα στο στρατό πριν από κάποιες δεκαετίες. Σήμερα παρατηρούμε έτσι ότι υπάρχει ανάγκη συνένωσης και κοινή χρήση για να παρέχονται οι δυνατότητες που απαιτούνται ε, και όπως είπε ο κ. Γκάλες ε, υπάρχει αυτή η απέτηση ηγεσία ε, και προς εκεί κινούνται οι πολιτικές, οι πολιτικές. Δεν είμαστε αυτός σκοπός από όλες τις απόψεις. Από την άποψη λοιπόν των στρατιωτικών πόρων είναι προτιμότερη η καλύτερη χρήση αυτών των εξαιρετικά μειωμένων πόρων όπως έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Από αυτή την άποψη η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων όπως είπε ο κ. Ε, Ρένεμαν ε, στο πλαίσιο μιας διεθνούς δύναμης διάσωσης, ό,τι και αν την ονομάσουμε, αυτή θα ήταν μια μόνιμη, δεν θα ήταν μια μόνιμη, δηλαδή θα είναι ουσιαστικά μια δύναμη εφεδρείας και οι φορολογούμενοι σίγουρα θέλουν οτιδήποτε υπάρχει να χρησιμοποιείται στο μέγιστο δυνατόν και όσο το δυνατόν συχνότερα. Ένα πλεονέκτημα μιας τέτοιας δύναμης είναι η δυνατότητα προσαρμογής, η ευελιξία και η μια οργάνωση με διευκολυντές που μπορούν να επιτελέσουν πολλαπλές εργασίες. Εμείς ε, θα βρισκόμαστε εκεί για να προσφέρουμε αρρωγή ως αντίδραση στις κρίσεις. Λόγω αυτών των δυνατοτήτων θα μπορούμε να πάμε στα πιο δύσκολα μέρη και σίγουρα εμείς δεν θα είμαστε εκείνοι που θα διορθώσουμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα ε, μίλησε η κυρία Λέζιν για την ΑΕΤ. Ε, ήταν πριν από το σχηματισμό της υπηρεσίας ε, εξωτερικής δράσης και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης πρέπει να μπορεί να παρέχει ολική, ολικό αποτέλεσμα. Εμείς συμβάλλουμε σε πολλούς τομείς, είμαστε Είμαστε πολύ λίγοι στρατιωτικοί μεταξύ των ε, υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ μικρό κομμάτι και αυτό που τονίζουμε είναι ότι θέλουμε να συνεργαστούμε. Ανέφερε η κυρία Νέτση ανησυχίες για το πώς η στρατιωτική δομή αλληλεπιδρά με άλλους φορείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πραγματική ανησυχία της μεροληψίας ε, και τις διατήρησης της ημεροληψίας ε, οργανισμών όπως της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ. Τα παίρνουμε όλα αυτά πολύ στα σοβαρά και συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν και ειδικότερα την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ για να υποστηρίξουμε με όποιον τρόπο μπορούμε χωρίς να βλάψουμε την, την αμεροληψία. Από αυτή την άποψη συνεργαζόμαστε στενά με το Κεντρό Συντονισμού βοηθάμε σε στρατηγικές διαδικασίες και άλλες προσπάθειες και έτσι έχουμε μια διαρκή συνεργασία με τη Γενική Διευθύνση ΕΚΟ που υπάρχει εδώ και κάποιο καιρό αυτή η συνεργασία και συνεχίζεται μέσα στη νέα εποχή της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Και οι κατευθυντήριες γραμμές του Όσουλ εφαρμόζονται σε αυτά τα θέματα. Άλλες ερωτήσεις ο κύριος Τάνεκ, συγγνώμη ανέφερε το ζήτημα για το κέρος της Αφρικής. Πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα όπου ο στρατός βοηθά άμεσα τη διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής όσον αφορά το λοιμό. Ο λόγος που έφτασαν με ασφάλεια τα εμπορεύματα του Διεθνούς Επιστημιστικού Οργανισμού χωρίς ε, να επηρεαστούν από την πειρατεία ήταν το αποτέλεσμα της επιχειρήσης Αταλάντα που έχει εκδιπλωθεί στι ε, σομαλικές ακτές ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια αυτών των ζωτικών ε, αποστολών. Με 100% επιτυχία μέχρι σήμερα, όχι μόνο επιτυχία, αλλά και που εξασφάλισε την προστασία, τη συνεχή προστασία όταν ε, ε, επιδεινώθηκε ο λοιμός. Αυτά με οδηγούν στο ζήτημα που ανέφερε ο πρόεδρος. Αυτή η τελευταία σας ερώτηση κατά πόσο, πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Είμαστε πιο ενωμένοι από ό,τι παλιότερα. Εγώ το πιστεύω. Αποκτά και μεγαλύτερη σημασία η συνεργασία μεταξύ μας λόγω του pooling and sharing και δεδομένου του γεγονότος ότι είμαστε πολύ λιγότεροι από ό,τι παλιότερα. Είναι επίσης σημαντικό διότι η επιπτώση της κλιματικής αλλαγής ε, για όλο και μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζει πιο άμεσα όλο και περισσότερους ανθρώπους. Μόνο τα τελευταία χρόνια πόσα περιστατικά οδήγησαν σε εμπλοκή του στρατού σε όλο και μεγαλύτερη έκταση για παροχή των πρώτων βοηθειών που βοήθησαν, διευκόλυναν εκείνων που έπρεπε να πάρουν τη σκητάλη τη αρρωγή στη συνέχεια. Ελπίζω έτσι να απάντησα μερικέ από τι σημαντικέ ερωτήσει που τέθηκαν από του διάφορου συμμετέχοντε. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ κύριο Μπχέο. Ευχαριστώ. Απλώ θα ήθελα να μιλήσω για το πολύ είναι sharing και για την σημασία της κατάρτισης. Εκεί είναι πολύ σημαντική η συνεργασία του στρατιωτικού με του πολιτικού σκέλους. Και θα πρέπει εδώ να έχουμε κοινέ προδιαγραφές, κοινού κανόνες μεταξύ ημών και ημών, για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε όλες αυτές τις καταστάσεις στην Ευρώπη πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σπένσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι ήθελα να κάνω έκκληση στα μέλη να μην ασχολούνται με τον τίτλο, αλλά με την ουσία της έκθεσης. Όταν εγώ ήμουν πρόεδρος στην Επιτροπή ΦΕΤ, ένα από τα λιγότερο ελκυστικά πράγματα που είχα να κάνω είναι να διαπραγματεύομαι με τις άλλες επιτροπές όταν έπρεπε να μοιραστούμε κάτι. Η συνεργαστία είναι σημαντική αλλά ο τίτλος θα πρέπει να αλλάξει δεδομένου ότι για πιο άλλο θέμα ε, μιλούμε ως συστηματικό θέμα. Τέλος πάντων, πολύ καλά ήταν τα σχόλια και της, και της Επιτροπής και του εισηγητού. Θα πρέπει να δούμε Όπως φαίνεται σε έναν ε, ε, πίνακα που έχουμε εμείς στο Foreign Office, με, αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα και αν δεν κάναμε σωστό σχεδιασμό, με τι θα έμοιαζε ένας τέταρτος κόσμος που θα γεννιότανε. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της ασφάλειας. Μία συνάδελφος ε, είπε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάζους μπέλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάζους μπέλη εδώ στην Ευρώπη, αλλά ήδη στις χώρες της Ασιατικές, πρέπει να πω ότι υπάρχει σχεδόν πόλεμος, κατάσταση πολέμου στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Κινέας. και νομίζω ότι το θέμα της παροχής ύδατος μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικό πόλεμο. Δεύτερον, η εμπειρία μου όταν έχω να κάνω με ε, αξιωματίουχους υψηλού επίπεδου είναι ότι το τελευταίο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν είναι η κλιματική αλλαγή. Δεδομένου ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται όλα τα θέματα ασφαλείας που έχουν στο επίπεδό τους. Στη ΣΥΠΑ το θέμα αυτό πραγματικά είναι μια καυτή πατάτα στα χέρια των πολιτικών. Αλλά πολλοί έχουν δει περί τίνος πρόκειται, ξέρουν το πρόβλημα, θέλουν να το συζητήσουν και με άλλους στρατιωτικούς και νομίζω ότι θα πρέπει με διαφάνεια και ανοιχτό πνεύμα και με όλους να συζητήσουμε αυτό το θέμα και τους Βραζιλιάνους και με τους ε, Ρώσους και με τους Κινέζους και να δούμε εφόσον επηρεάζει όλες τις κοινωνίες μας πώς θα μπορέσουμε να χειριστούμε αυτό το θέμα. Οι Βρετανοί και οι ε, οι Γερμανοί είπαν ότι θα πρέπει να γίνεται ετησίω μια διάσκεψη για να ασχολούμεθα με τα θέματα αυτά όλοι. Τώρα, αυτού του τετάρτου βαθμού χάρτης όπως σας λέω που έχουμε στο Foreign Office. Αυτός ο χάρτης. Όπως είπε και ένας ε, συντηρητικός συνάδελφος, θα πω το εξής. Δεν έχει σημασία που είστε πλέον όταν μιλούμε για το τι ε, προκάλεσε την κλιματική αλλαγή. Συνέβη. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μπορεί του πάντε και την Ινδία και την Κίνα και τον Καναδά και όλο τον κόσμο και την Ιαπωνία να του επηρεάσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και βεβαίως αυτό ήταν κάτι το οποίο οι ίδιοι οι Βρετανοί το ήξεραν και δεν ασχολήθηκαν. Πέρασαν στο επόμενο βήμα. Πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα. διότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, ε, θέμα το οποίο να πρέπει να ασχοληθούμε και να μην αφήσουμε τα πράγματα να επιδεινωθούν, διότι θα καταλήξουμε σε καταστροφή. Θα πρέπει επίσης να δούμε για αυτό το θέμα πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι συζητήσεις που γίνονται από, σε πολιτικό επίπεδο. Κάπου νομίζω ότι χάσαμε το στόχο και δεν θα πρέπει να αφήσουμε την στρατιωτική διάσταση στο περιθώριο. Πρόκειται, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Η εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει εφόσον είναι οργανωμένη, να ηγηθούν όλων αυτή η στρατηγική θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχαστεί και ο ρόλος και η διάσταση στρατηγική. Αυτά ήθελα να πω στους αδέλφους. Κοιτάτε την ουσία. Τροπο, ε, πι, κάντε τροπολογίες επί της ουσίας αυτή την έκθεση. Ο τίτλος είναι άλλο θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει. Και θα πρέπει να δείτε επίσης και μακροχρόνια ποια πολιτική και στρατηγική θα αναπτύξουμε. Όχι μόνο κοντόφθαλμα για πέντε χρόνια, τα επόμενα 10, είκοσι και παραπάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, ε, πλούσια. Και κύριε Ταράντ, έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε εσείς οριστικά τη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μετέχοντες και οφείλω να ομολογήσω το εξής. Στην αρχή πρέπει να πω δεν ήμουν χρήσιμη ε, για το κατά πόσον το σχέδιο της εκθεσής μου ήταν χρήσιμο. Εσείς όλοι με πείσατε ότι πράγματι τελικά παρουσίασα μια πολύ χρήσιμη έκθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ λακωνικό το συμπέρασμά σας, αλλά και χρήσιμο θα έλεγα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τους ε, προσκεκλημένους μας και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης που αφορά σε έκθεση πρωτοβουλίας από τον κύριο Τούνε Κέλαμ σχετικά με την ασφάλεια ε, στον κυβερνοχώρο και στην άμυνα. Θα περιμένουμε λιγάκι. we continue, but it's to to to ask. Uh, dear colleagues, I would like to ask to continue discussions maybe. Αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως τις ιδιωτικές σας συζητήσεις μπορείτε να τις κάνετε λίγο αργότερα ή έξω από την αίθουσα. Λοιπόν, έχουμε την έκθεση για την ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και χώρες ε, όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, μεγάλες αλλά και μικρές, αλλά εξίσου σημαντικές, όπως η Εσθονία παραδείγματος χάρη, έχουν υποφέρει από επιθέσεις ε, στον κυβέρνοχώρο. Γιατί τέτοιου είδου επιθέσεις ε, μπορούν να διαταράξουν την υποδομή ή ε, να καταστήσουν παντελώς ανεποτελεσματικές τις στρατιωτικές μας δυνάμεις. Ίσως λοιπόν μπορεί ο κύριος Κέλαμ να μας εξηγήσει πώς ακριβώς μπορούμε να προστατευτούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ίσως ε, είναι συμβολικό το γεγονός ότι η κυβερνοασφάλεια υπολείπεται ακόμα, γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις ε, φυσικές καταστροφές. Δεν μπορούν να επηρεάσουν την ε, καθημερινότητά μας, αλλά οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται μυστικά οι περισσότεροι πολίτες ε, δεν τις ε, συνειδητοποιούν, δεν ενημερώνονται ούτε καν από τους ε, ηθήνοντες, από δημοσίους υπαλλήλου σε υψηλά κλιμάκια. Παρ' αυτά, στην έκθεση αυτή, με την έκθεση αυτή, καλό όλους τους αρμόδιους να θεσπίσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα κυβερνοασφάλειας ένα σύστημα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχει μια ε, κατάλληλη στρατηγική. Ήρθα σε επαφή με διάφορους ε, εταίρους, με εκπροσώπους μας, δικούς μας στο, ΝΑΤΟ, σε υπηρεσίες άμυνας και η έκθεσή μου διαιρείται σε εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Άμυνας σε δραστηριότητες ε, ΣΔΙΤ σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα κάνω τώρα και ορισμένες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασίας να ε, παρισφρήσει το στοιχείο της κυβερνοασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δραστηριότητες ε, και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε αυτή την ανάγκη, γιατί αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όλα αυτά έχουν σχέση και με την ποικιλομορφία των απειλών, γιατί δεν πρόκειται μόνο για το ότι μπλοκάρονται τα συστήματα ενημέρωσης, αλλά μπλοκάρεται και η υποδομή μιας χώρας, κάτι που σημαίνει ότι παραλύουν σημαντικά συστήματα υποδομής, παραλύουν ολόκληρα κράτη. Το βασικό λοιπόν θέμα είναι να υπάρχει καλύτερος συντονισμός ε, και ε, καλύτερη συνοχή και συνέπεια. Όσον αφορά τώρα σε μία από τις τελευταίες εξελίξεις, είχαμε μία θετική εξέλιξη, την εξέλιξη του Μαΐου αυτού του έτους, όπου όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησαν ομάδες, υπεύθυνε ομάδες, ε, για να ανταποκριθούν σε έκτακτες περιπτώσεις ε, που θα αφορούν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτές λοιπόν οι ομάδες ε, θα προσφέρουν βοήθεια έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δυναμικό κυβερνοάμυνας. Ο ρόλος αυτών των, ε, της του Ευρωπαϊκού Φορέα, όπως ε, ξέρετε, είναι και να εμβαθύνει τη συνεργασία του με τον ΝΑΤΟ. Ένας λοιπόν από, ένα από τα θέματα που μας απασχολούν είναι ότι μόνο ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ε, δαπανά 2% των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη αυτό τομέα και πέντε κράτη δεν έχουν προβλέψει κανένα κονδύλι για αυτή την έρευνα και την ανάπτυξη, τουλάχιστον αυτό ε, συνέβαινε πριν από δύο χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τα κρατημέλη να διοχετεύσουν κονδύλια και να επενδύσουν σε ε, συλλογικές δραστηριότητες ε, έρευνας ε, και ασφάλειας, κυρίως όσον αφορά στην κυβερνοασφάλεια. Όσον αφορά τώρα στα κράτη-μέλη, το πρώτο καθήκον είναι να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν την κυβερνοασφαλειά τους και την στρατηγική τους και αυτό μάλιστα αμελητή. γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ε, βελτιώσει πολύ το να υπάρχει και ένας ε, πρακτικός οδηγός για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Εξάλλου, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ορίσουν στις στρατιωτικές τους δυνάμεις ε, που έχουν και ειδικέ τέτοιες μονάδες κυβερνοασφάλειας. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχουν μηχανισμοί συνεργασίας έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Προτείνουμε λοιπόν να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο υποχρεωτικής ε, συνεργασίας και ανταλλαγής ε, πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, και κάτι άλλο που αφορά στα κράτη-μέλη, να αναπτύξουν δικά τους προγράμματα έκτακτης ανάγκης, όπου συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων και αυτά κάτω από το πρίσμα της ανάλυσης κινδύνων. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με το ότι πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή εκπαίδευση. Σωστή εκπαίδευση για όλους τους υπαλλήλους δημόσιων φορέων. Αν υπήρχε αυτό, θα είχαμε μια μεγαλύτερη βοήθεια. Πάντω, ε, σε γενικές γραμμές θα έλεγα, απευθυνόμαστε στα κράτη-μέλη και τα καλούμε να διασφαλίζουν μια υγιεινή, αν θέλετε, στον κυβερνοχώρο, να υπάρχει προστασία, να μπορούν να παρεμποδίζουν την εμφάνιση κινδύνων. Κατά τη γνώμη μας, αυτό σημαίνει να υπάρχει σωστή εκπαίδευση για την κυβερνοασφάλεια στα σχολεία, στα σχολικά προγράμματα και αυτό από, την, όσο, από μικρή ηλικία. Όσον αφορά τώρα την, ε, το δημόσιο φορέα, αυτό που είναι σημαντικό είναι να ενθαρρυνθεί καταρχήν ο ιδιωτικό τομέα που είναι υπεύθυνο για τι περισσότερε δραστηριότητε που αναπτύσσονται στον χώρο, να ενθαρρυνθεί να περιλαμβάνει ε, διαχείριση κρίσεων και για άλλη μια φορά ακούσαμε όλοι ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει η σωστή εκπαίδευση ε, για όλους τους υπαλλήλους. Όσον αφορά τώρα στη διεθνή συνεργασία, νομίζω ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης οφείλει να λειτουργήσει ε, προληπτικά όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και να προσπαθήσει τα στοιχεία αυτής να τα συμπεριλάβει σε όλες τις δραστηριότητες. Βεβαίως όλα αυτά σχέδια, ε, συσχετίζονται και με την ολοκλήρωση μιας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας. Όμως ε, όλα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως πρόφαση για να αποφεύγει κανείς ε, την αντιμετώπιση τέτοιου προβλημάτων στις σχέσεις του με τρίτες χώρες. Εμείς λοιπόν έχουμε υποβάλει ένα ερώτημα σε πάρα πολλά επίπεδα κατά πόσον η σύμβαση της Βουδαπέστης ε, αρκεί τι ακριβώς ε, χρειαζόμαστε, μήπως ε, χρειαζόμαστε ένα νέο επίπεδο, μια νέα νομική βάση και ίσως και νέες απαντήσεις. Αλλά μέχρι τώρα οι απαντήσεις που υπάρχουν είναι ότι η σύμβαση της Βουδαπέστης είναι ένα ικανοποιητικό εργαλείο. Εκείνο που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα, διότι έχουμε κατά νου να προχωρήσουμε σε υψηλότερο επίπεδο, είναι να τροποποιηθεί η σύμβαση της ε, Λισαβόνας από όλα τα κράτη-μέλη. Και επίσης ε, οι διεθνείς μας ε, εταίροι να παραμένουν πιστοί να τηρούν αυτή τη σύμβαση. Πάντως, το άμεσο καθήκον για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και για τα κράτη-μέλη είναι να επιδιώξουν μια ευρύτερη διεθνή συμφωνία για ε, θέματα συμπεριφοράς, ε, για καλές ε, πρακτικές στον κυβερνοχώρο. Αυτό λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το να υπάρχουν και ελάχιστες προδιαγραφές, ε, ελάχιστοι όροι για το πώς μπορεί κανείς ε, να προλάβει τις ε, κυβερνοεπιθέσεις. Ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο κυβερνοχώρος δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο αρνητικά. Η ελευθερία ενημέρωσης που προσφέρει ο κυβερνοχώρος, οι δυνατότητες που υπάρχουν διασύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για τη δημοκρατία και την ελευθερία όπως το διαπιστώσαμε στην περίπτωση των αραβικών επαναστάσεων αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να έχουμε κατά νου και αυτό το τόσο ε, θετικό στοιχείο. Όσον αφορά τώρα στις σχέσεις με το ΝΑΤΟ, νομίζω ότι μία βασική προσέγγιση ε, η βασική προσέγγιση θα πρέπει να είναι και περιεκτική. Δεν μπορούμε απλά να επαναλαμβάνουμε αυτά που κάνει το ΝΑΤΟ. Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά και πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να έχουμε μια συνεπέστερη προσέγγιση είναι το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε στο εξής δίλημα κατά πόσον η επίθεση στον κυβερνοχώρο είναι η καλύτερη μορφή άμυνας. Έχουμε κατά νου τον ιό που προσέβαλε τα ε, συστήματα αεροπορικών ε, πτήσεων. Ε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη διάδοση τέτοιου είδους ειδών. Πρέπει να ζητήσουμε καλύτερες απαντήσεις. Επίσης, σε περίπτωση ε, κυβερνοεπιθέσεων πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα καταφύγουμε στις ρήτρε αλληλεγγύης ε, τόσο με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας όσο και στους κόλπους ε, του ΝΑΤΟ όπου τα περισσότερα κράτη-μέλη είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα, οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να προκαλέσουν τεράστια ζημιά μπορεί να συγκριθεί η ζημιά αυτή με φυσική επίθεση. Σε περίπτωση φυσική σωματικής επίθεσης μπορούμε να επικαλεστούμε την ε, ρήτρα αλληλεγγύης. Αλλά σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο αυτό δεν είναι τόσο σίγουρο. Βεβαίως ε, πρέπει να συνεργαστούμε με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες στον τομέα αυτό. Πριν από δύο χρόνια η ομάδα εργασίας ε, για την κυβερνοασφάλεια και το κυβερνοέγκλημα ε, εισήχθη και τον Μάιο κατά την τελευταία μας συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Πολιτειών, συζητήσαμε εκ νέου το θέμα αυτό. Σε γενικές λοιπόν γραμμές ε, θέλω να πω ότι αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για το ότι έλαβαν υπόψη τους αυτό το πρώτο σχέδιο. Ε, βασίζομαι στη συνεργασία σας ε, και στις ε, τροπολογίες που θα καταθέσετε και ευτυχώς έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας διότι η καταληκτική μερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 6η Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ εμείς, σκιώδης εισηγητές, συντάκτης. Κύριο Γιάννη από του Σοσιαλδημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη διότι έφτασα κάπως αργά. Γιατί ήμουν σε άλλη επιτροπή. Θα ήθελα να πω το εξή. Δεν χρειάζεται ίσως να τονίσω και αν χρειάζεται το κάνω. Πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση η οποία με μεγάλη σοβαρότητα συνετάχθη από τον εισηγητή. Πρόκειται για ένα θέμα γενικά καινούριο και για το ευρύ και για τους επαγγελματίες και για τους πολιτικούς. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε παιδαγωγικό έργο μονίμως για να κατανοήσουν όλοι πόσο η μεγάλη σημασία πρέπει να προσδώσουμε στην κυβερνοάμυνα και στην κυβερνοασφάλεια η έννοια αυτή ούτως ή άλλως όπως ξέρουμε είναι καινούρια και δύσκολη. Και πρέπει να δούμε ποια θα είναι η έννοια που θα γίνει γενικά αποδεκτή, διότι υπάρχουν διαφορές. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο κίνδυνος που ενέχει για κάποιους το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, ενημέρωσης, επικοινωνίας. και την διπλή χρήση την οποία μπορεί να κάνει κανείς στον τομέα αυτών των τεχνολογιών εις βάρος της άμυνας και της ασφάλειας. Πώς θα μπορέσουμε να βρούμε τα κατάλληλα όπλα λοιπόν για να πολεμήσουμε την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτή της έκθεσης είναι ότι σημαίνει ότι το θέμα αυτό δεν είναι στατικό. Το θέμα εξελίσσεται οποιαδήποτε τροπολογία ή οποιαδήποτε, οποιοδήποτε μέτρο προστασίας πάρουμε, επειδή εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα τα πράγματα, μπορεί να εμφανιστεί ως ξεπερασμένο σε κάποιους μήνες. Κατά την άποψή μου, πάρα πολύ ορθά λοιπόν ο εισηγητής αναφέρει διάφορα επίπεδα συνεργασίας εντός κάθε κράτος μέλους, δεδομένου ότι είναι πολύ διαφορετική η νομοθεσία και οι κανόνες που ισχύουν εντός κάθε χώρας, συνεργαστεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των διαφορετικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, στην διεθνή κοινότητα, μέσω υπηρεσιών και οργανισμών των οποίων είμαστε και μέλη. Το ΝΑΤΟ, Φερρυπίν, ο ΙΕ, με τις οργανώσεις του. Ούτως ή άλλως πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα έχει στις πολιτικές συζητήσεις όλο και περισσότερη σημασία και θα αποτελέσει και τον πυρήνα του οράματος που θα έχουμε εμείς για το θέμα αυτό και των απόψεων που θα αναπτύξουμε. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό το Κοινοβούλιο νομίζω ότι του προσδίδει την ε, σημασία που του αξίζει. Δεν έχουμε προβλήματα, υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές για τις οποίες θα καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε καμία ουσιώδη διαφορά Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω στην αίθουσα εκπροσώπους των Φιλελευθέρων και των Πρασίνων, ενώ σκιώδης. Ε, κύριε Λόζινγκ, λοιπόν, μπορείτε να μιλήσετε. Κοιτάξτε, λέει η κυρία Λόζινγκ, δεν χρειάζεται να αναφερθώ στη σημασία του διαδικτύου και στη σημασία που μπορεί να έχει η διατάραξη αυτών των συστημάτων επιπτώσεις τους ε, στη ζωή μας. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε σε βάθος πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς και νομίζω ότι και ο εισηγητής το είπε αυτό, υπάρχει συνεργασία με τον ΝΑΤΟ υπάρχει και η επίκληση ε, της ε, περίπτωσης ε, επίθεσης σε μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα, σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει άμυνα ή αντεπίθεση με στρατιωτικά μέσα. Ποιον θα πυροβολήσουμε, τι θα γίνει. Σήμερα το πρωί Πραγματικά δεν κατάλαβα, δεν το πίστευα σχεδόν ότι τους ε, πειρατές ε, πρέπει να τους ε, πλησιάζουν μόνο στρατιωτικά σκάφη και όχι αλλιευτικά. Αυτά όλα που λέγονται εδώ, εγώ τα βρίσκω ανοησίες. Νομίζω ότι οι ειδικοί για υπολογιστές πρέπει να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια του διαδικτύου. Μόνο έτσι μπορούμε να προστατευτούμε. Αυτά όσον αφορά την άμυνα. Και υπάρχει βέβαια και μια άλλη διάσταση του θέματος, το θέμα της ε, επίθεσης. Αναφέρθηκε ότι στην ε, Bundeswehr, στο στρατό της ε, Γερμανίας, εκπαιδεύεται μια ειδική ομάδα ε, που θα είναι ειδική για κυβερνοεπιθέσεις. Αυτή υποτίθεται θα συνεργάζεται με τις Ηνωμένε Πολιτείε και το ΝΑΤΟ. Αυτή η επιθετική διάσταση, τι ακριβώς είναι, νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε και να το σκεφτούμε. Δηλαδή, αν μερικοί χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ως όπλο, Αυτά που λέγονται βέβαια δεν είναι φαντασιώσεις, γίνεται κάτι τέτοιο. Αν ισχύει αυτό, τότε πρέπει και εγώ να διερωτηθώ κατά πόσον όλα αυτά που συζητώνται εμπίπτουν στο κεφάλαιο έλεγχος των εξοπλισμών. Γιατί αν στο μέλλον το διαδίκτυο λάβει στρατιωτική μορφή, τότε αυτή όλη η τεχνολογία του διαδικτύου εμπίπτει στις εξαγωγές εξοπλισμών. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί αυτό ο εισηγητής, γιατί εγώ δεν βλέπω να το θίγει στην έκθεσή του. Πάρα πολύ ωραία, τιξατε πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ο κύριος Τερχόφ από την ομάδα των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον εισηγητή. Πολύ σωστά ο κύριος εισηγητής ε, καταδεικνύει τη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και ειδικότερα για την καταπολέμηση νέων κινδύνων. Επίσης ε, αναφέρει ότι χρειαζόμαστε επίσης εθνικές στρατηγικές διότι εκεί υπάρχουν οι περισσότερες δυνατότητες και οι περισσότερες υποδομές και το ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε υποδομές σε εκείνο το επίπεδο πιστεύω ότι είναι πολύ καλό που καταδεικνύει ο εισηγητής το ενδεχόμενο δημόσιας, ε, δημόσιων και ιδιωτικών ε, ε, συνεργασιών σε αυτόν τον τομέα. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Πολύ δουλειά πρέπει να γίνει στον ιδιωτικό τομέα και είναι εξαιρετικά δύσκολο να ζητήσουμε από το δημόσιο τομέα να ασχοληθεί με ορισμένα από αυτά τα ζητήματα. Επίση, πιστεύω είναι πολύ ενθαρρυντικό που μιλάει ο εισηγητή και για τις καλέ πλευρές του διαδικτύου. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη διάδοση σωστών δημοκρατικών πρακτικών και την καταπολέμηση δικτατορικών καθεστώτων. Μια άλλη καλή πτυχή είναι το γεγονό ότι ο εισηγητή αναφέρει πω ε, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξουν τα δικά του συστήματα και τις δικές τους πλατφόρμες ασφάλειας ε, διαδικτύου. Ο εισηγητής λοιπόν πιστεύω έχει συμπεριλάβει πολύ σημαντικά ζητήματα στην έκθεσή του με ευρεία ε, οπτική. Είναι πολύ θετική αυτή η έκθεση, ωστόσο θέλω να επισημάνω ότι και οι δυνατότητες των κρατών μελών όσον αφορά τις δομές είναι σημαντικό να συντονιστούν. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν χρειαζόμαστε κάποιο νέο διεθνή οργανισμό για να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την πολιτική ομάδα του ECR. Ο κύριος Κάμπελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εκθέση αυτή πιστεύω είναι εξαιρετικά σημαντική για ένα πολύ σημαντικό τομέα. Αποτελεί τεράστια απειλή σήμερα που μας επηρεάζει όλους σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα. Πρόσφατα υπήρξε μια έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα σας πω από ποια εταιρεία. Μια εταιρεία έχασε εκατομμύρια λιρών λόγω επίθεσης κυβερνοεπίθεσης. Πιστεύω ότι κλιμακώνεται ουσιαστικά η απειλή. Γίνεται όλο και πιο σοβαρή. Έχω δύο ερωτήσει. Αυτό που δεν κατάλαβα δεν, κανείς δεν διατίθεται θεραπεία ακριβώ από που προέρχονται αυτές οι επιθέσεις. Γνωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες, τις έχουμε στην κατοχή μας, μπορούμε να είμαστε σαφείς όσον αφορά την προέλευση Υπάρχουν υποψίες, υπόνοιες για την Κίνα, για τη Ρωσία, για κάποιους οργανισμούς μυστικούς, ε, συνηθισή ύποπτη φυσικά. Γιατί είμαστε τόσο ευγενικοί. Είναι γιατί δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι προέρχονται από εκεί ή απλά γνωρίζουμε από πού έρχονται αλλά δεν θέλουμε να το συζητήσουμε. Το δεύτερο σημείο και είναι αρκετά ενδιαφέρον για να λειτουργήσουν, για να έχουν αποτέλεσμα αυτέ οι επιθέσει να μα δημιουργήσουν πρόβλημα, χρειάζεται αρκετά μεγάλη υποδομή τόσο για την προετοιμασία των επιθέσεων όσο και για την εξαπολύσή του. Φυσικά, μόλι εξαπολύθουν αυτέ οι επιθέσει, πόσο αυξημένα είναι αυτά τα δίκτυα αυτοί οι οργανισμοί. Όλα αυτά είναι νέα, δεν ξέρω ακριβώς τι ορολογία να χρησιμοποιήσω. Πόσο ανεπτυγμένες είναι οι δυνατότητες υπεράσπιση μας όσον αφορά τους ιούς. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλον ένα σκιωδή εισηγητή, τον κύριο Τάραντο, ε, από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μοναδική αυτή η ευκαιρία να μιλάει ο εισηγητής στη γλώσσα μου. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν και εγώ τα αισθονικά. Οι πράσινοι στο κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που κυκλοφόρησε μια τέτοια έκθεση στην Επιτροπή μας. Παρότι οι χώρες έχουν σύνορα και έχουν επιτύχει την ανεξαρτησία τους, την κυριαρχία τους δεν συμβαίνει το ίδιο στον κυβερνοχώρο. Εκεί τα σύνορα δεν είναι σαφή. Ο ορισμός μιας επίθεσης πρέπει να είναι πολύ σαφής ο ορισμός της λέξης επίθεσης ότι, ώστε όλοι να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς αποτελεί επίθεση. Διότι όπως γνωρίζουμε η Εστονία είναι μία από τις χώρες που έχει ήδη βιώσει κύβερνο επίθεση. Δεύτερον, στο όσον αφορά αυτή την έκθεση. Θα θέλαμε να καλυφθούν ζητήματα όπως ε, πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση αυτών των τομέων. Αυτά ήθελα να επισημάνω προς τη στιγμή. Αφού παρουσιαστεί η έκθεση θα υποβάλουμε και τροπολογίες εφόσον καταστεί απαραίτητο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συγητή, τον συναδελφό μας, τον κύριο Κάλαμ, για την έκθεση αυτή. Για τις ε, συγκεκριμένες προοπτικές δράσεις που προτείνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών, για την διασύνδεση που θα πρέπει να γίνει σε διεθνές επίπεδο και κυρίως με τους εταίρους, τους ε, ε, πολύ σημαντικούς για μας, το ΝΑΤΟ και τη ΕΠΑ. Και επίση για την δυνατότητα συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εγώ ήμουν από αυτούς που συμμετείχαν στις συζητήσεις που είχαμε με τους Αμερικανούς συναδέλφου τον τελευταίο Μάιο στην Κοπενχάγη και Πρέπει να πω ότι συζητήσαμε αυτό το θέμα σε μια ειδική συνάντηση και όπως όλα τα άτομα τα οποία αρχίζει να καταλαβαίνει τι σημαίνει στο χώρο του, στο κυβερνοχώρο, πραγματικό, πραγματικά ανησύχησα. Και είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί και σε επίπεδο των κρατών μας, των πολιτών μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για, θέλω να κάνουμε κάτι για την ε, άμυνά μας. Έχουμε να κάνουμε για κάτι το οποίο μπορεί ε, το οποίο έχει ισχύει παγκοσμίω, ξεπερνάει τα σύνορα, δεν γνωρίζει σύνορα. Άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε αν αποτελεσματικά το όλο θέμα. Το ορόσημο μεταξύ εσωτερικής, αν θέλετε, εθνικής ή εξωτερικής ασφάλειας σχεδόν δεν υπάρχει. Πρέπει να πω ότι επίσης ήμουν σε μία συνάντηση που έγινε όπου ακούστηκαν τα διάφορα μέτρα για την κύβερνοασφάλεια, μία συνάντηση με την Ευρωπόλο, που είναι ε, πάρα πολύ ε, σημαντικός οργανισμός που ασχολείται με αυτά τα θέματα και όπως ξέρουμε αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο σημαντικό έργα υποδομής. Άρα δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε τη σημασία του. Και στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκή Ένωσης θα πρέπει να έχουμε μία συνεκτική πολιτική και χρηματοδότηση ώστε να αναπτύξουμε αυτή τη στρατηγική για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις κυβερνοεπιθέσεις. Ή στα πλαίσια της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ή για την καταπολέμηση της εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρέπει, όπως λέει ο συνάδελφος Κέλλαμ, να επιστήσει την προσοχή μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών και της ε, ισορροπίας που πρέπει να επιτευχθεί. Για να μην ε, ανοίξουμε ε, τις πόρτες αν θέλετε και τα παράθυρα ορθάνυχτα, δεδομένου ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο από κάποιες χώρες και αναφέρομαι κυρίως σε κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής. Επίσης, ε, εδώ αναφέρεται η ρήτρα της αλληλεγγύης, αν υπάρχει μια σοβαρή επίθεση κατά μιας χώρας τη Ευρωπαϊκή Ένωση. όπως συνέβη και στην Εστονία. Είδαμε ότι κάτι τέτοιο λοιπόν μπορεί να συμβεί και ξέρουμε ότι εδώ μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο ε, πάρα πολύ σημαντικά έργα υποδομής σε όλες τις χώρες μέλη. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτά τα κέντρα Επικοινωνίες. Δεν ξέρω εάν θα μπορέσουν ε, να γίνουν αυτά τα οποία λέγονται ε, για τη δημιουργία αυτών των κέντρων στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν μπορούν να είναι ε, λειτουργικά αυτά τα κέντρα, τα εθνικά και κέντρα αριστείας προβλέπονται. Δεν ξέρω αν έχουν δοθεί κατάλληλοι πόροι από διάφορε χώρε και πρέπει βεβαίω να παραδεχτούμε ότι η οικονομική κρίση έχει τρομερά αρνητικέ επιπτώσεις στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε μέχρι να εγκριθεί εξής τι ακριβώς έχει γίνει και σε επίπεδο και των μελών και σε επίπεδο επιτροπής. Θα ήθελα επίσης να τονίσω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Πρόκειται για ένα από τα θέματα που συζητήσαμε με τους Αμερικανούς συναδέλφους και με τους πραγματογνώμονες και είδαμε ότι όντως υπάρχει μεγάλη δυσπιστία μεταξύ τους και υπάρχουν πάρα πολλά συμβάντα τα οποία δεν καταγράφονται, τα οποία δεν αναφέρονται διότι πολλές φορές ο ιδιωτικός τομέας ε, επιλέγει να τα αποκρύψει, πράγμα το οποίο έχει καταστροφικές συνέπειες στο όλο σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποιες ρυθμίσεις και κάποια θέματα να είναι υποχρεωτικά. Μετά την κατάρτιση να υπάρχει κάποια υποχρέωση για όλους. Από τη στιγμή την οποία μιλούμε, και όχι μόνο μιλούμε, έχουμε να κάνουμε με αυτά τα δεδομένα που είναι στο Dropbox. Κανένας δεν λέει πλέον τίποτε. Μπορούν όλα τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί εκεί να καταστραφούν με ένα κλικ. Πράγμα καταστροφικό για κράτη, για δημόσιες διοικήσεις, για επιχειρήσεις και δεν υπάρχουν κανόνες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επενδύσουμε και στον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίσουμε τα προβλήματα και τις απειλές και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, σε θέματα διεθνούς συνεργασίας, κυρίως με το ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ. Είναι πολύ εύστοχα τα σχόλια που περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή, αλλά δεν θα πρέπει να μην παραγνωρίσουμε και κάποιες δράσεις που αναλαμβάνουν οι συνομιλητές μας στη ΣΥΠΑ. Ε, από πού προέρχονται όλες αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις, τι ελέγχθη για την Εστονία, ίσως από την Κίνα, από την Εστονία, από τη, συγγνώμη, από την ε, Ρωσία. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία επίσης που, που διάβασα στο New York Times, ε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι πολύ ανησυχητικά και μπορούν να πολλαπλασιάσουν την, ε, τα πυρηνικά, τους πυρηνικούς οπλισμούς ε, ανά τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί για να μην ανοίξουμε το κουνδί της πανδώρας που θα είναι καταστροφικό για όλους μας. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι λέχτησαν τα περισσότερα και κατέστη σαφές ε, πόσο ευρύ είναι το θέμα. Η μόνη δυσκολία που υπάρχει είναι να ε, συγκεντρώσουμε τις απόψεις διότι είναι δυνατόν σε αυτό το θέμα στην ε, κυβερνοασφάλεια μπορεί να θίγονται μεμονωμένοι πολίτες ε, πολλοί μπορούν ε, να υποστούν συνέπειες να παραλύσει το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να θυγούν και ε, στρατιωτικές μονάδες, οποιοδήποτε. Πάντως, όσον αφορά το δικό μας τον τομέα, ο οποίος έχει σχέση με ευαίσθητους δημόσιους φορείς και όπου αντιμετωπίζουμε από κοινού την απειλή, ως ε, θεσμοί Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Να δούμε τι είδου ε, μηχανισμοί άμυνας υπάρχουν, όπου ο καθένας πρέπει να εγκαθιστά μόνος του αυτούς τους ε, μηχανισμούς ασφαλείας και η υπεραξία προκύπτει από το συντονισμό που λαμβάνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, ε, ο συνάδελφος ε, μας επισήμανε ε, πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Όσον αφορά τώρα στο ερώτημα το οποίο έθιξε προηγουμένως η συνάδελφο, δηλαδή πώς θα πρέπει κανείς στρατιωτικά να αντιδράσει σε κυβερνοεπιθέσεις. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν τίθεται έτσι το ερώτημα κυρίως αν δεν γνωρίζουμε από ποιον προέρχεται η επίθεση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο το ΝΑΤΟ, προς το παρόν τουλάχιστον, λέει ότι η κυβερνοεπίθεση δεν οδηγεί στην επίκληση του άρθρου 5. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς το άρθρο 5 λόγω κυβερνοεπίθεσης. Αυτή είναι η πολιτική στάση του ΝΑΤΟ. Ίσως αυτό να αλλάξει. Ε, Παραδείγματο χάρη, αν μπορεί να αποδειχτεί από ποιον προέρχεται η επίθεση. αν ας πούμε τεθούν εκτός λειτουργίας ιδιαίτερα ευαίσθητες υποδομές ή αν τεθεί σε κίνδυνο η ζωή ανθρώπων ή αν χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να έχαν τη ζωή τους ε, παλαιότερα οι άνθρωποι με όχι τόσο καθαρά εισαγωγικά μέσα στο πεδίο της μάχης. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Όμως, θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα και αντίστροφα. Δηλαδή, αν προέρθει κυβερνοεπίθεση από στρατιωτική πηγή, θα είναι δυνατόν η απάντηση να είναι επίσης στρατιωτική. Θα είναι δυνατόν να ξεκινήσει πόλεμο στο διαδίκτυο. Όλα αυτά είναι θέματα ιδιαίτερα δυσάρεστα αλλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί όλο και περισσότερο μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι που κανείς μας ε, δεν τους επιθυμεί αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δυνατόν να ασκείται πίεση με αυτό τον τρόπο και βία βέβαια ε, και όχι όπως γινόταν ε, τους προηγούμενους αιώνες. Εμείς ως δημοκρατικά ε, σταθερά κράτη, σίγουρα δεν είμαστε εκείνοι ε, που σκεφτόμαστε με όρους επίθεσης, αλλά περισσότερο με όρους άμυνας, το πώς θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Όμως, όπως είναι γνωστό, για να χορέψουν ταγκό πρέπει να υπάρχουν πάντα δύο. Εάν λοιπόν εντοπίσουμε ότι υπάρχει, ε, υπάρχουν τέτοιου είδους πιθανότητες, θα πρέπει και εμείς να σκεφτούμε πώς θα αντιδράσουμε. Θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλέ ε, τεχνικές δυνατότητε αντίδραση. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω τίποτα άλλο επ' αυτού. Ε, το καθήκον μας είναι όχι να βρούμε λύση επί παντός του επιστήτου, αλλά να επισημαίνουμε στην εκτελεστική εξουσία, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει πρόβλημα, αυτή είναι η κατάσταση αντικειμενικά και παρακαλούμε αναζητήστε λύσεις. Δεν είναι δουλειά του Κοινοβουλίου να προσφέρει πάντα τις λύσεις. Η εκτελεστική εξουσία πρέπει να το κάνει αυτό. Και η έκθεσή μας αυτό το σκοπό έχει. Ευχαριστούμε. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας, αλλά έχουμε κάποια χρονικούς περιορισμούς. Παρακαλώ λοιπόν είστε σύντομοι. Κυρία Βαλερία Νοβάλη, της Γενικής Διεύθυνσης Connect. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Εκ μέρου τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα ήθελα να χειρισώ και σημειώνουμε αυτή την ε, έκθεση της Επιτροπής Άμυνας και Ασφαλές. Έχουμε πολλά, πολλούς ανησυχίες δεδομένου ότι αυξάνονται οι απειλές ταχύτατα γεγονό που θέτει σε κίνδυνο την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Ειδικότερα διότι η κοινωνία βασίζεται στον κυβερνοχώρο σε μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι κατά την Κομισιόν δεν μιλάμε μόνο για περιστατικά εγκληματικής φύσης, μπορεί να υπάρξουν επίσης και φυσικές καταστροφές και τεχνικά λάθη που να οδηγήσουν σε προβλήματα. Επίσης, η Κομισιόν συμφωνεί με το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφερόμενοι στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ειδικότερα οι δυνατότητες ε, ε, στα κράτη-μέλη είναι αρκετά νομιογενείς. Επίσης, συμμεριζόμαστε την άποψη ότι Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών, ιδιωτών ενδιαφερομένων. Είναι όντω το ζήτημα παγκόσμιας φύσης και πρέπει να αντιμετωπιστεί μαζί με τους διεθνείς μα εταίρους. Επίσης, λοιπόν, θεωρούμε ότι αυτή η έκθεση είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Πράγματι, η Κομισιόν και η ΠΑΤΕΚ εκπρόσωπος ε, ε, συνεργάζονται για να παρουσιάσουν ε, στο φέτος την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στρατηγική αυτή θα αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος που να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες, τις βασικές αξίες. Αυτή η στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, ειδικότερα δράσεις βελτίωσης της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών. Επιπλέον η Επιτροπή θα προτείνει ένα νομοθετικό μέσο ώστε να δώσει κίνητρα στα κράτη-μέλη για να αναπτύξουν τις εθνικές τους δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα. Ρωτώντας, ε, ζητώντας για παράδειγμα το προσδιορισμό των αρμόδιων αρχών στον τομέα, την υιοθέτηση εθνικών στρατηγικών ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, ε, την σύσταση ομάδων ε, ανταπόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. καθώς και την έγκριση σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης στο νομοθετικό μέσο. Αυτό προτείνει και ένα πλαίσιο για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μέλων στον τομέα της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών. Θα προτείνουμε κάποιες απαιτήσει για τον ιδιωτικό τομέα, για ενδιαφορμένους κλειδιά του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα πρέπει να υιοθετήσουν κατάλληλα μέτρα επικινδυνότητας, να αντιμετωπίσουν τα, συστήματα, τα προβλήματα στα συστήματα και να αναφέρουν τα περιστατικά ασφαλείας που επηρεάζουν σημαντικά την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Αυτό θα συνεπάγεται την παροχή πληροφοριών από τον ιδιωτικό τομέα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των οικονομικών. Στον αφορά τη στρατηγική για την ασφαλεία των δικτύων, θα αντιμετωπίζετε τα ζητήματα ασφαλείας με την πρόταση δράσεων, για να δοθούν κίνητρα στον τομέα τεχνολογικών πληροφοριών και επικοινωνιών για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας σε αυτόν τον τομέα και των επενδύσεων. Επίσης θα προτείνει δράσεις, ευαισθητοποίηση σε διάφορα επίπεδα από τους πολίτες μέχρι τους ε, υπαλλήλου έως και σε πολιτικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση Όσον αφορά την επικινδυνότητα, η στρατηγική αυτή επίσης θα αφορά δράσεις ενίσχυσης της καταπολέμησης του κυβερνού εγκλήματο. Θα προτείνει δράσεις ανάπτυξης ε, συνεκτικών ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της διεθνούς διάσταση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και για την προώθηση της ε, δυνατότητας δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες. Η στρατηγική επίσης θα αφορά τις πτυχές υπεράσπισης στον κυβερνοχώρο, άμυνα στον κυβερνοχώρο όσον αφορά ειδικότερα τις συνέργειες μεταξύ μη στρατιωτικών και στρατιωτικών ε, υποδομών ασφαλείας στο διαδίκτυο. Ε, τέλος, ε, θα αντιμετωπίζει τις πτυχές διακυβέρνησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ευθύνες σε θέματα ε, ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και στη διασάφηση αυτών των ευθυνών. Ε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι λοιπόν με αυτή την πολύ επίκαιρη έκθεση και σημειώνουμε τις δράσεις ε, που θα χρησιμεύσουν ως πληροφορία για αυτό το έργο, για αυτή τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό το σημείο σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Επανήλθε ο κύριος Φρανκ. Του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, η έκθεση αυτή είναι για μας μια ενθάρρυνση για την συνεχιζόμενη εργασία την οποία επιτελούμε για την κυβερνοστρατηγική σε επίπεδο επιτροπής με τη συνεργασία των συναδέλφων. Η Επιτροπή ασχολείται με αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια. Αλλά αυτό το οποίο έλειπε μέχρι τώρα είναι η κάλυψη, κάτι από την οποία θα έχουμε όλα αυτά τα θέματα, μια στέγη δηλαδή όλων των προσπαθειών κοινή. Σήμερα πρέπει να γίνει αυτό, δεδομένου ότι η στρατηγική αυτή έχει σχέση με την νομοθετική δράση που έχει αναλάβει η Επιτροπή. Και βεβαίω έχουμε χρονοδιάγραμμα το οποίο μάλλον πρέπει να πούμε ως σε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε έτοιμοι το τρίτο τρίμηνο και θέλουμε να έχουμε χειριστεί πολλά σημαντικά θέματα μέχρι τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και η συνάδελφο, ε, της Επιτροπής σας και η συνάδελφος της Επιτροπής σας εξήγησε τι ακριβώς θα κάνει και η, υπηρεσία εξωτερική, εξωτερικής συνεργασίας της Επιτροπής Συμβουλίου θέλουμε εμείς να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι να εξασφαλίσουμε ασφαλείς συνθήκες πρόσβασης στον κυβέρνο χώρο, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα όλων των χρηστών και να προσπαθεύσουμε τους πάντες από κυβερνοεπιθέσεις για να επιτύχουμε μεταξύ άλλων και οικονομική ανάπτυξη. μιλούμε ρησό για κάποιες διαφορές μεταξύ της ε, κυβερνοελευθερίας και της ε, προστασίας του κυβερνοχώρου από επιθέσεις. Αλλά ο στόχος μας είναι η προστασία του κυβερνοχώρου. Θα ήθελα να πω πόσο σημαντική είναι η συζήτηση που γίνεται για τις ε, τους κανόνες και τις προδιαγραφές που πρέπει να υπάρχουν στον τομέα αυτό εκ μέρου των κρατών μελών. Αυτό είναι κάτι το οποίο στη δικασία άρχισε πέρσι με τη διάσκεψη του Λονδίνου και θα συνεχιστεί εφέτος με δεύτερη διάσκεψη στην Βουδαπέστη και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε εκεί να παρουσιάσουμε μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να καταδεικνύει ποια είναι η προσέγγιση μας. Δύο λόγια τώρα για την κύβερνο άμυνα. Επιλαμβανόμεθα και αυτή της ε, πτυχής του προβλήματος μαζί με τους συναδέλφους του στρατιωτικού σκέλους. Είμαστε επίσης ε, και σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και ακόμη κάτι να προσθέσω Η διάσκεψη της Βουδαπέστης, βασισμένη στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, για μας είναι ο κύριος αντικειμενικός στόχος για να δημορφώσει πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποτελέσει την βάση συνεργασίας με τρίτες χώρες για να προστατευτούμε από κυβερνοεπιθέσεις. Αναφέρθηκε Επίσης όσον αφορά τις τρίτες χώρες, στενή συνεργασία την οποία έχουμε στο ομάδα εργασίας με τη ΣΥΠΑ, που ασχολείται με διάφορα σχετικά θέματα. Θα έχουμε επίσης συνεργασία και μετά από συζητήσει με την Ινδία για θέματα πολιτικού διαλόγου για την ασφάλεια θα δούμε το Σεπτέμβριο πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την Ινδία καθώς και μελετούμε με ποιες άλλες χώρες θα κάνουμε παρεμφερή διάλογο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπριά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυο λόγια για να συμπληρώσω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ασμπέκ από την εξωτερική υπηρεσία. Πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη η έκθεση αυτή, δεδομένου ότι τώρα θέλουμε στον τομέα της κυβερνοασφάλειας να καταρτήσουμε την πολιτική μας ευρωπαϊκό επίπεδο. Είδαμε ποια είναι η θέση των κρατών μελών Καταρχάς τώρα με εμά είναι πολύ πιο ανοιχτοί, θέλουν να χειριστούμε από κοινού αυτό το θέμα. Το θεωρούν προτεραιότητα σε σχέση με το τι σκέφτονταν πέρσι, αλλά σε πολλές χώρες ακόμη δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Τι θέλουν να κάνουν μόνοι τους, θέλουν να κάνουν σε θέματα περιορισμένη συνεργασία με άλλες χώρες και τι θέλουν να κάνουν σφαιρικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι πάρα... και θα πρέπει να γίνει, διότι θα πρέπει να ξέρουμε στο μέλλον στο επίπεδο της δικής μας οργάνωσης άμυνας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια θέματα μπορούμε να χειριστούμε από κοινού. Για να δείξω πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Όπως ξέρετε, ασχολούμαι πάρα πολύ με τα σφακέλους που αφορούν τον ε, ενιαίο ε, ευρωπαϊκό ουρανό. Τα θέματα των δικτύων και στο στρατιωτικό σκέλος και στο πολιτικό σκέλος της αεροπορίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μερικά χρόνια όλα τα αεροπλάνα θα κινούνται βάσει ε, της σύνδεσής τους με αυτά τα δίκτυα και θέλουμε να είναι σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας όσοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ε, αρχίζουμε να συνεργαζόμαστε από τώρα και να απτύξουμε συστήματα για να είναι ασφαλείς οι πολίτες μας σε λίγα χρόνια. Επίση υπάρχει και ανθρώπινος παράγοντας ουσιαστικής σημασίας. Και κάποιες συμπεριφορές θα πρέπει να αλλάξουν. Όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι η κυβερνοασφάλεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα λοιπόν δίνω και πάλι το λόγο στον εισηγητή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θετικά σας σχόλια και για τις συμβουλές που μου δώσατε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο μόλις τώρα είπε ο συνάδελφός μας από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ισχύει πράγματι αναζητούμε μία μορφή ε, και είναι σημαντικό ε, να ξέρουμε τι δεν αφορά αυτή η έκθεση. Αυτή η έκθεση δεν αναφέρεται στο διαδίκτυο. Υπάρχει μια έκθεση για επιθέσεις ανάμεσα σε συστήματα, κρίσιμα συστήματα πληροφορικής. Και επίσης δεν αναφερόμεθα στο ΝΑΤΟ ή πώς να δώσουμε απαντήσεις σε στρατιωτικές επιθέσεις ε, τέτοιου είδους. Αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στο να προετοιμάσουμε το πολιτικό έδαφος για να επεκτείνουμε την ευαισθητοποίησή μας ή τις ε, δυνατότητες ε, που κρύβει μια κυβερνοεπίθεση. Εδώ πρόκειται για μια πολύ σοβαρή απειλή. και εξακολουθεί να επικρατεί η άποψη ότι έχουμε καθυστερήσει. Δεύτερον, μπορούμε πολιτικά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και εμπειρίες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα, αλλά τα κράτη-μέλη δεν είναι στον ίδιο βαθμό προετοιμασμένα. Είναι τεράστια διαφορά στην προετοιμασία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συντονισμός. Και το τρίτο καθήκον μας είναι η εκπαίδευση στην κυβερνοϊγιεινή. Ε, αυτό μοιάζει να είναι πρωτόγονο που σας λέω, αλλά επειδή επισκέφτηκα το Εστονικό Κέντρο Αριστείας για την Κυβερνοασφάλεια, εξεπλάγει με το πώς ε, ενθαρρυνθήκαμε να ασχοληθούμε με αυτό το βασικό πρόβλημα της ε, κυβερνοεκπαίδευσης. Τώρα, ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά, για αυτές τις επιθέσεις, ποιος είναι υπεύθυνο. Ακούσαμε τον εμπειρογνώμονά μας και έγιναν και προτάσεις ε, προς τη Ρωσία την Κίνα ως τις ε, βασικές πηγές ε, κυβερνοεγκληματικών δραστηριοτήτων. Ε, Βεβαίω ε, δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε τέτοιου είδους υπενιγμούς στην έκθεσή μας. Εκείνο που είναι προφανές είναι ότι σε αυτόν τον τομέα υπάρχει ένα είδος αρνητικών συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή ακόμα και τα κράτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδιώτες ε, που μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν και να χρησιμοποιούνται με την ε, ιδιωτική τους ιδιότητα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο να <clears throat> προσφέρουμε κίνητρα σε αυτούς που το επιθυμούν να κάνουν κάποια καλή δουλειά, να ε, προσφέρουν πρωτοβουλίες να διασφαλίζουν τις δικές μας τις ε, κυβερνοδιασυνδέσεις. Η ρήτρα αλληλεγγύης αναφέρθηκε στην παράγραφο υπαριθμών 3 της έκθεσης. Για άλλη μια φορά λοιπόν απευθύνομαι στην Επιτροπή καλώντας την να εξετάσει το κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρχει επίκληση αυτής της ρήτρα σχετικά με την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, σε τελική ανάλυση είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις ελευθερίες και τους περιορισμούς. Αυτή είναι η βασική δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαίρομαι που συμφωνούν με αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε κι εμείς ε, με τη δική μας την ταπεινή συνεισφορά σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Και άλλη μια φορά να σας πω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Δεν μπορούμε να τα ότι, μπορούμε, ότι έχουμε χρόνο και ότι μπορούμε συνεχώς να αναβάλουμε τα προβλήματα. Το βασικότερο θέμα είναι η συνεργασία. Είμαστε πρόθυμοι όλα αυτά να τα επεξεργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι αν ε, η πρόκληση αυτή ε, το δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο εγγύς μέλλον με θετική έκβαση. Ευχαριστούμε. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτό το σημείο, το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης η δεύτερη εξέταση ενό σχεδίου νομοθετικής γνωμοδότησης αφορά την πρόταση της Κομισιόν για κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθιερώνει στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικής Ασφάλειας, το Ταμείο για την χρηματοδοτική στήριξη για τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις. Δίνω λοιπόν το λόγο στον στην εισηγήτρια, την κυρία Ελέν Φλότρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα ξανά την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις δικές μου τροπολογίες για αυτό το νομοσχέδιο που έτσι δημιουργεί ένα υπόβαθρο για τις θεωρήσεις και για τα σύνορα ξεκινώντας από ένα πιο γενικό υπόβαθρο για την εσωτερική ασφάλιση σας υπενθυμίζω πολύ γρήγορα τα κυριότερα σημεία αυτών των τροπολογιών οι οποίες είναι 55 τον αριθμό περίπου το πρώτο σημείο για τη συνοχή των ενωσιακών πολιτικών κυρίως με χρωσό της έκκλησης της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης δεύτερον για να συμπεριληφθούν οι επαρκείς αναφορές σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων κυρίως η συμμόρφωση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης με το ε, κοινωτικό κεκτημένο να ληφθούν υπόψη τα πολυβέστα ζητήματα του ασύλου στα σύνορα αφήνοντα τα ζητήματα για το άλλο μέσο τα ζητήματα του ασύλου και της μετανάστευσης που δεν, στο άλλο μέσο που δεν περιλαμβάνεται εδώ στη συνέχεια πολλές τροπολογίες που αφορούν τη σχέση μεταξύ της πολιτικής θεωρήσεων και της κινητικότητας και τέλος πολλές επαναλαμβανόμενες τροπολογίες ε, που θα μπορούσαμε ενδεχομένως να ψηφίσουμε μαζικά μία για αντικατάσταση και το είχαμε συζητήσει με την Κομισιόν και συμφωνούσε η έννοια του νόμιμου ταξιδιού ήταν λίγο αφηρημένη και δεν αναφέρεται στα τρέχοντα έγγραφα της Ένωσης, συνεπώς θα πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι πιο ε, γνωστό οργάνωση και διευκόλυνση της τακτικής μετανάστευσης. Στη συνέχεια θα αντικαταστήσουμε το ζήτημα των απειλών με εκείνο της επικινδυνότητας και τις προκλήσεις όπως, είναι όπως πρότεινε η κυρία Κοπά. Εκεί η κυρία Κοπά θα παρουσιάσει τις δικές της τροπολογίες που είναι 14, ο κ. Κάζα έχει υποβάλει 3, αυτοί έχουμε 10 Επτά τροπολογίε βάσει όλων αυτών. Έχουμε πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών στο Στρασβούργο με επτά συμβιβασμούς στο, η πλειοψηφία τους ενσωματώνουν τις προτάσεις της κυρίας Κοπά εξαλλού επειδή μπορέσαμε να υπολογίσουμε ότι για την συγκίτρια του ΕΛΚΑ υπήρχαν δυσκολίες, συμφωνίες ε, για ορισμένους συμβιβασμούς. Είναι πως μετά από αυτή τη συνεδρία των σχεδόν πρότεινα τροποποιήσεις που ελπίζω θα βοηθήσουν να έχουμε την υποστήριξή της. Κυρίως όσον αφορά την συμβιβαστική τρία εκεί αντικατέστησα το Through Principle of Solidarity and Fair Sharing με Following the Principle of Solidarity and Fair Sharing Επίσης προτείνω, μετά από συμφωνία με την κυρία Κοπά, να καταργήσουμε την αναφορά στο burden sharing που είχε προβλήματα για την κυρία Βέντερε. Συμβιβαστική 4 λοιπόν, γνωρίζοντας ότι η συμβιβαστική 3 αναφέρεται σε αυτό το θέμα και ότι το άρθρο 80 της συνθήκης ε, αναφέρεται ρητά. Μετά από πρόταση της κυρίας Κοπά, η αντικατάσταση ε, της απειλής με επικινδυνότητα κίνδυνο θα γίνει όταν ε, θα γίνεται εφόσον εννοείται επικινδυνότητα ή με πρόκληση εφόσον ε, σε τουλάχιστον δύο σημεία του κειμένου, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Το πρώτο σημείο νομίζω είναι η τροπολογία 63 της κυρίας Κόπα και θα αποσύρω την τροπολογία μου εκεί όπου προτείνω ρίσκα και πρότεινα μια τροπολογία για τη δική μου τροπολογία 8 ώστε να συμπεριληφθεί αυτό το ζήτημα του challenges, δηλαδή προκλήσεις. Στη συνέχεια... Η κυρία Κοπάρα θα σας παρουσιάσει τις αλλαγές που επιθυμεί αυτή. Όσον αφορά τις τροπολογίες του κύριου Κάζα, είναι εδώ ο κύριος Κάζα. Όχι, επειδή ήθελα να του ζητήσω διευκρινήσεις. Ε, υπάρχει κάπως πρόβλημα, όπως φαίνεται, το να προσθέσουμε ένα συνεκτικό μηχανισμό μεταξύ των δύο μέσων. Μπορούμε να το πούμε, αλλά ούτως ή άλλως διασφαλίζεται ήδη από το γεγονός ότι υπάρχουν γενικές διατάξεις στο σύνολο των μέσων που διασφαλίζουν τον παραλληλισμό των μεταρρυθμίσεων μεταξύ του μέσου συνόρων και θεωρήσεων και του ασύλου και μετανάστευση. Μπορούμε να το πούμε βέβαια αν το επιθυμεί ο κύριος Κάζα. Και μετά όσον αφορά την τροπολογία 64, 62 και 64 θα ήθελα να το συζητήσω μαζί του διότι μπορούμε ενδεχομένως να αποδεχθούμε τουλάχιστον ένα κομμάτι των δύο τροπολογιών αυτών για τις υπόλοιπε τροπολογίες επτά δεν θα συμπεριληφθούν στη συμβιβαστική υπέβαλε 14 η κυρία Κοπά. Εγώ προτείνω να υποστηρίξουμε τι τροπολογίες τη κυρία Κοπά που ουσιαστικά αφορούν βελτίωση του κειμένου, κυρίως όσον αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις, αναφορές σε κείμενα που έχουν ήδη υιοθετηθεί, ώστε να υπάρχει συνοχή με κυρίως τον κανονισμό Frontex και την καθολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας. Αυτές οι τροπολογίες μου φαίνεται ότι εμπλουτίζουν το κείμενο, γι' αυτό λοιπόν τι υποστηρίζω. Thank you. ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον του ΕΛΚ. Εσείς θα τον αντικαταστήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώ η συνάλφο που ασχολείται με το θέμα δεν μπόρεσε να έρθει. Γι' αυτό θα μιλήσω εγώ σύντομα και θα είμαι πολύ σύντομο. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, της ΕΛΚ ε, συμφωνούσαμε απόλυτα με την πρόταση της Επιτροπής και γι' αυτό το λόγο δεν συμφωνούσαμε με τις αλλαγές της ε, κυρίας Φλότρ. Τώρα, οι συμβαστικές προτάσεις της κυρίας Κοπά πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη διατύπωση και την ουσία. Βέβαια, παρόλα αυτά, εμείς, αν κάνουμε τη σύγκριση, βρίσκουμε καλύτερες τις προτάσεις της Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν το ΕΛΚ θα κάνει το εξής. Στο 2 θα συμφωνήσουμε. Ε, κατά τα άλλα, θα απορρίψουμε τις ε, άλλες τροπολογίες οι συμβαστικέ προτάσει. έτσι κι αλλιώ προέκυψαν χωρί εμά. Και το πώς θα ψηφίσουμε στην τελική ψηφορία, αυτό θα το συζητήσουμε ακόμα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί. Η κυρία Κοπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ ε, τον εισηγητή για τη δουλειά μας και να πω ότι στηρίζω τις συμβαστικές ε, προτάσεις που είναι ισορροπημένες. Νομίζω ότι παρά τις ε, αντιρρήσεις και επιφυλάξεις που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των ε, ε, σκιωδών εισηγητών, ίσως ε, το ΕΛΚΑ αναθεωρήσει τη θέση του και συμφωνήσει ή έστω συζητήσει για κάποιες εξ αυτών. Γιατί είπανε ξεκάθαρα ότι στηρίζουν τη θέση της Κομισιόν. Όμως είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί αν διαφωνούν, ας πούμε, με την συμβαστική 2, Τρία διορθώνει η κυρία Κοπά. Με συγχωρείτε, έκανα εγώ λάθος που βασίζεται στις ε, πρόνοιες της ε, συνθήκης και ε, την πέντε, όπου γίνεται μόνο αναφορά των ονομάτων των συνθήκων και των συμφωνιών. Κάτι το οποίο όλοι μας συμβόμαστε. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή το σκεπτικό πίσω από την απόφαση να μην στηρίξουν τις τροπολογίες αυτές. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εμείς δεν είχαμε βασικές, βασικά προβλήματα με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση της είναι θετική, βασίζεται στην αλληλεγγύη και στον επιμερισμό των ευθυνών ε, και γίνεται σχέση ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια. Όμως, Θέλουμε να αλλάξουμε λιγάκι το πώς παρουσιάζεται όλο αυτό το θέμα, να προβάλλουμε περισσότερο το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, όπως επίσης ε, και να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ε, παροχής υπηρεσιών ε, σε ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν για επιχειρηματικούς λόγους. Νομίζω έτσι πήρατε μια γενική εικόνα των ε, τροπολογιών μου, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω και ορισμένα θέματα που είναι περισσότερο τεχνική φύσεω. Την 70 ή 17 μάλλον, με συγχωρείτε. Εκεί αναφέρομαι σε διορθωτικέ ε, πράξει, διότι δεν θα ήθελα να υπάρξουν περιπτώσει όπου η ε, Επιτροπή καταθέτει ε, μέτρα ανακατανομή κονδυλίων προσθέτοντας κόστος που δεν καλύπτεται. Τώρα, για να διασφαλιστεί ότι το εθνικό πρόγραμμα στη τελική ανάλυση θα αποδώσει, θα πρέπει οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Και επιπλέον αποδίδω μεγάλη σημασία στην βελτίωση των δυνατοτήτων ε, και σε συμφωνία με την εισηγήτρια θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όταν γίνεται αναφορά στο κόστος προσωπικού, εδώ περιλαμβάνεται και το κόστος της εκπαίδευσης, παράρτημα 3. Και τέλος, κάτι που συμφωνήσαμε και συζητήσαμε, είναι να χρησιμοποιούνται σωστά οι όροι απειλές και προκλήσεις στο κείμενο. Είχαμε μια συζήτηση επ' αυτού, όπως είπε και η κυρία Φλότρ εξάλλου, η απειλή κατανοώ πολύ καλά ότι έχει μια αρνητική απόχρωση. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε πού ακριβώς θα χρησιμοποιούμε τη λέξη κίνδυνος και πού ακριβώς τη λέξη πρόκληση. Και όπως ε, είπε και η κυρία Φλότρ, θα διευκρινίσει περισσότερο το θέμα των τροπολογιών. Την ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή της. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε. Ο υπάρχει σχέδιο εισηγητής από το Άλντε, δεν βλέπω κάποιον, ούτε από το ΙΣΕΑΡ. Κυρία Λέζινγκ, λοιπόν. Gut, langsam geht mir die Stimme aus für... Βέβαια, πρέπει να σα πω ότι σιγά σιγά αρχίζω να χάνω τη φωνή μου, βραχνιάζω, γιατί εγώ σήμερα είμαι εδώ σκιώδη ηγητρία για τα πάντα, επί παντό του επιστητού. Τέσσερις ε, λοιπόν οι τροπολογίες της ε, κυρίας Κοπά συμφωνώ ε, στη σωστή κατεύθυνση είναι για να επιφέρουν ελάφρυνση. Επίσης όσον αφορά την διαδικασία σύλλου συμφωνώ πρέπει να διεκπαιρώνει τη διαδικασία αυτή με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτά είναι σημαντικά θέματα για τους ανθρώπους. Εμείς βέβαια έχουμε άλλα βασικά προβλήματα με τη Frontex. Εδώ γίνεται μια θετική αναφορά επ' αυτών. Και ε, έχουμε μεγαλύτερα ουσιαστικά προβλήματα με την πρόταση της ε, Επιτροπής με την κατεύθυνση που ακολουθεί αυτή η πρόταση. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι μέχρι σήμερα δεν καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα. Ε, Παραδείγματο χάρη δεν καταλαβαίνω αυτό το σημείο στην πρόταση που αναφέρεται με σαφήνεια και γίνεται λόγος για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως global player, παγκόσμιος παίκτη, ε, ότι θα έχει μία επιρροή μόχλευσης. Τώρα, τι είδου ε, επιπτώσεις θα προκύψουν, αυτά μέχρι σήμερα δεν τα έχω καταλάβει. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει από τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να εξετάσουμε το θέμα και νομίζω όλα τα άλλα ε, θα πειράσουν βέβαια το πώς θα ψηφίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Η κυρία Φλότρ. Τα σχολιά σας, κυρία Φλότρ. Ναι. Για να απαντήσω στον κύριο Γκάλερ, ο οποίος... Ε, για συγγνώμη, μια στιγμή, με συγχωρείτε. Ίσως έκανα λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Οντουάν Σαβαρή, αναπληρωτή ε, μονάδα. Είναι παρόν. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προτάσεις και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Είμαι πάρα πολύ σύντομες, διότι και εγώ τις ανακαλύπτω τώρα αυτές τις ε, τροπολογίες συμβαστικές. Θα είναι δύσκολο, λοιπόν, αυτή τη στιγμή να αποφανθεί η Επιτροπή. Εκ πρώτης όψεως υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο να δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Τούτο λεχθέντος, θα πρέπει να μελετήσουμε περαιτέρω την διατύπωση κάποιων τροπολογιών μετά από αυτή την ε, πρώτη ματιά που έριξα. Εμείς βεβαίως δεν θα Ε, κάνουμε τίποτε πριν να συζητηθεί σε δικό σας και να συμφωνηθεί σε δικό σας επίπεδο από το φθινόπωρο και μετά θα έχετε την επίσημη απόψή μας. Ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι βρήκα ότι δεν είναι και τόσο πολύ ευγενικά σαν τα πει ο κύριο Γκάλης για πολλούς λόγους. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς συμβιβαστικές ε, να βρίσκει συμβαστικές λύσεις όταν δεν έχει διάφορες τροπολογίες. Η συνάδελφό σα, η σκέδωση συγγήτρια, ξέρει πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Συζήτησα μαζί της όλα αυτά τα θέματα και τις τροπολογίες και εξ ονόματός μου τις δύο προτάσεις που έκανα εγώ λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που συζητήσαμε στο Στρασβούργο να τα μεταφέρετε στην κυρία Βέντερε. Διότι εσείς εδώ επαναλάβετε τη θέση της ε, θέση που μας είχε εκφράσει στο Στρασβούργο. Μας είπε ότι συμφωνεί με τη συμβαστική πρόταση 2 και εσείς το ίδιο επαναλάβατε. Εγώ λοιπόν πρέπει να πω ότι δεν έχω πολλά στοιχεία στη θέση μου για να κάνω συμβαστικές προτάσεις και τροπολογίες και δεν διαφωνείτε φαντάζομαι με αυτά τα οποία λέω. Πολύ καλά, σας ευχαριστώ. Πιστεύω λοιπόν Έχουμε ολοκληρώσει την ημερήσια διάταξη και μπορούμε να διακόψουμε εδώ τη συνεδρίασή μας και φυσικά θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιστές να μείνουν και τον κύριο Ντανζάν, ο κύριος τη ο πρόεδρος της Επιτροπής, θα έρθει.